Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε. Καθίστε παρακαλώ. ξεκινάμε σήμερα το πρωί με μια κοινή συνεδρίαση των επιτροπών ΛΥΜΠΕ και φεμ για την εμπορία ανθρώπων. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Εύα Μπρίτς Βένσον, τη συνάδελφη από την Επιτροπή Γυναικών. Να σας υπενθυμίσω περί τίνος πρόκειται. Τον προηγούμενο Μάρτιο είχαμε μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εμπορία ανθρώπων και την κατάργηση της απόφασης πλαίσιο 2002 Επειδή το θέμα της εμπορίας ανθρώπων είναι αρμοδιότητα τόσο της Επιτροπής Γυναικών όσο και της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, αποφασίστηκε ότι με βάση τον άρθρο 51 του κανονισμού του Κοινοβουλίου θα κάνουμε κοινή συνεδρίαση. η νομοθετική διαδικασία επί τη βάση της πρότασης της Επιτροπής συνεχίζεται. Στις 10 Ιουνίου είχαμε και ένα σεμινάριο επί του θέματος. Και η Άννα Χέτ από την Επιτροπή μας και η Edith Bauer από την Επιτροπή Γυναικών θα παρουσιάσουν τις εκθέσεις τους. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι 22 Ιουλίου το μεσημέρι και στις 2 Σεπτεμβρίου θα γίνει η συνεδρίαση. Θα δώσω το λόγο τώρα στις συνεισηγήτριες. Η κυρία Χέντ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους όσους ε, κάνανε μια εξαιρετική εργασία για αυτήν την ε, πρόταση για την σωματεμπορία την ε, κυρία Μπάουερ, την ε, Κλάουδια από τη Γραμματεία της ΛΥΜΠΕ και τη Φαμπρίσια από την Επιτροπή Γυναικών. Εγώ και ε, ε κυρία Μπάουερ κάναμε μία κοινή πρόταση Πιστεύουμε ότι η συνεργασία για το άρθρο 51 λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και βασιστήκαμε στο ψήφισμα που παρουσιάσαμε τον Δεκέμβριο. Για μένα η πρόληψη είναι προτεραιότητα. και πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην πρόληψη όταν θα διατυπώσουμε την νομοθετική πρόταση. Πρέπει να σταματήσουμε τη ζήτηση της σωματεμπορίας. Η πρόταση ελπίζουμε ότι θα μειώσει τη ζήτηση και αυτό με ποινές πολύ πιο αυστηρές και επίσης κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Το τράφικινγκ θα πρέπει να γίνει πλέον κάτι το οποίο δεν θα ε, δίνει κέρδη ε, στο δίκτυο διακίνησης. Από 6 έως 12 χρόνια πρέπει να ανέβουν οι ποινές. Θα πρέπει επίσης ε, να υπάρχει δυνατότητα κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων των εγκληματιών ε, για να μπορέσουμε να αποζημιώνουμε τα θύματα. Χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία και βοήθεια στα θύματα, κυρίως ε, στα παιδιά. Πρέπει να παλεύουμε για το ε, των παιδιών. Τα θύματα της ε, σωματεμπορίας θα πρέπει να δικαιούνται δωρεάν νομικής βοήθειας και να έχουν και την ελευθερία να αποφασίζουν αν θα συμμετέχουν στην ε, ανακριτική διαδικασία ή όχι. Η βοήθεια προς τα θύματα είναι ένας ε, εύστοχος τρόπος ε, για να καταπολεμήσουμε το τράφικινγκ. Φυσικά χρειάζεται να έχουμε και μία προοπτική ως προς τα θέματα μετανάστευσης. Και αυτό για να καλύψουμε και πολίτες τρίτων χωρών που είναι θύματα της σωματεμπορίας. Επίσης ε, είπαμε και την αρχή της μη απέλασης, ε, της, ε, το, το no refoulement για τα θύματα της σωματεμπορίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία για τη συλλογή στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τα στοιχεία μαζεύονται στις διάφορες χώρες με διαφορετικούς τρόπους πληροφορίες ε, για το φύλλο, για την ηλικία, ε, ποιος ήταν ο στόχος ε, της σωματεμπορίας. Όλα αυτά θα πρέπει να μαζεύονται βάσει των δηλώσεων που γίνονται όπως επίσης θα πρέπει να καταγράφονται όσοι καταδικάζονται για σώματεμπορία όπως επίσης και οι ποινές που τους δίνονται. Λοιπόν, χρειάζεται ποινικοποίηση όλων αυτών των αδικημάτων και θα πρέπει να ξαναδούμε την ερμηνεία του άρθρου 15.4. Πρέπει να τιμωρούμε αυτούς που εκμεταλλεύονται ε, και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα θύματα της ε, σωματεμπορίας. Αυτό ευθυγραμμίζεται και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαγορεύει στους εργοδότες να απασχολούν θύματα σωματεμπορίας. Ευχαριστώ κυρία Μπάουαρ. Thank you so much. Uh, Ευχαριστώ. Τι να προσθέσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την πολύ αποτελεσματική συνεργασία αλλά και την Άννα για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε κάτι που δεν είναι σύνηθες υπό τον κανόνα 51 αλλά παρόλα αυτά λειτουργήσε τέλεια η συνεργασία. Τώρα, Ίσως θα μπορούσα να προσθέσω κάποιες απόψεις ή να πω κάποια πράγματα διαφορετικά. Το... Η εμπορία ανθρώπων έχει υψηλό προφίλ, μικρό, είναι, έχει υψηλό κίνδυνο αλλά μικρό προφίλ. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά δεν είναι αποτελεσματική. Πώς μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε τα πράγματα, να αυξήσουμε το κίνδυνο για όσους ε, επιδίδονται στην εμπορία ανθρώπων προκειμένου να τους αποτρέψουμε. Στις συζητήσεις με τη Europol μας είπαν ότι ότι αν δεν αλλάξει το περιβάλλον, αν δεν γίνει πιο αποτρεπτικό, θα παραμείνει αναποτελεσματική η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε ότι προκειμένου να προσανατολιστούμε περισσότερο προς τα θύματα, ίσως χρειάζεται να έχουμε αυστηρότερες κυρώσεις. Γι' αυτό επιστρέψαμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσθέσαμε ένα νέο τύπο κυρώσεων. Και αν, πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί δεν είχε γίνει και στο παρελθόν αυτό. Κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων όσων επιδίδονται στην εμπειρία ανθρώπων. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά ως αποτρεπτικό μέτρο. Το άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η αρχική νομοθεσία μιλούσε για τα θύματα από τρίτες χώρες. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά. Η αιτήσια εισρωή θυμάτων εμπορίας ανθρώπους είναι 70.000 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέφτουν θύματα της εμπορίας. Γιατί πλέον υπάρχουν χιλιάδες θύματα που προέρχονται από κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι αυτή η τυχή λοιπόν πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη. Μία άλλη νέα τάση είναι η εμπορία παιδιών και η εμπορία με στόχο την καταναγκαστική εργασία. Υπάρχουν λοιπόν ειδικέ διατάξεις που αναφέρονται σε αυτά τα δύο θέματα. Στο σχέδιο έκθεσης μιλάμε για έναν Ευρωπαίο συντονιστή. Θέλουμε οι εθνικοί συντονιστές να είναι ανεξάρτητα άτομα ή μηχανισμοί και έχουμε την εντύπωση, έχουμε πληροφορίες ότι αν δεν υπάρξει ένας Ευρωπαίος συντονιστής που θα συντονίζει τις διάφορες πολιτικές και θα συντονίζει αν θέλετε τους εθνικούς συντονιστές δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι αναπόφευκτη η χρήση του. Και υπάρχουν πληροφορίες από την Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθεί αυτή η θέση σε κάποια γενική διεύθυνση. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να είναι πιο υψηλή αυτή η θέση και να προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα καλό βήμα. Και σε σχέση με αυτό που είπε και η Άννα όσον αφορά μια ενιαία μεθοδολογία για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων. Υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές στο σχέδιο έκθεσης. Θα τα συζητήσουμε αυτά αργότερα, αλλά Νομίζω ότι αυτά που ανέφερα είναι οι βασικές αλλαγές τώρα με στόχο πάντα να κάνουμε πιο αποτελεσματική την νομοθεσία για τον τομέα αυτό. Και βεβαίως ε, αναμένουμε τη συζήτηση αλλά και τα σχόλια των συναδέλφων προκειμένου να βελτιώσουμε το σχέδιο έκθεσης. Και μία ερώτηση προσδοκώντας μια καλή συνεργασία με την Επιτροπή. και την Προεδρία. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την ανοιχτή συνεργασία που είχαμε και με τα δύο όργανα. Σε αυτή την πρόταση υπάρχει πρόθεση να ασχοληθούμε και με το θέμα της προσωρινής άδειας παραμονής. Θέλουμε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μελέτη εφαρμογής αυτής της οδηγίας αλλά να πω ότι έχουμε την εντύπωση ότι θα χρειαστεί αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Επιτροπή αν μπορούμε να βασιζόμαστε σε μία αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προσωρινή άδεια παραμονής, ενδεχομένως με διατάξεις για την προστασία μαρτύρων. Ευχαριστώ. Έχουμε 35 λεπτά και έχουν ζητήσει 7, 8, 9, 10 το λόγο. Θα ζητήσω από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σχολιάσουν πολύ σύντομα. Παρακαλώ, όχι παραπάνω από τρία λεπτά. Απλά τα βασικά. Μετά θα συνεχίσουμε με τη συζήτηση και στο τέλος θα ζητήσω από τις εισηγήτριες να συνοψίσουν. Πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τις 10 γιατί αναμένουμε τη Βελγική Προεδρία. Παρακαλώ λοιπόν δείξτε πειθαρχία. Καταρχάς ο κύριος Φλόρ εκ μέρους του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, σύντομος. Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτό το σχέδιο οδηγίας. Πρόκειται για ένα σχέδιο πολύ σημαντικό για όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο εργάστηκε ε, τόσο προσεκτικά και γρήγορα για αυτό το σχέδιο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και για την ε, λεπτομερή εκτενή εργασία των δύο εισηγητών που βελτιώνουν την πρόταση της Κομισιόν και για το Συμβούλιο και εμείς εργαστήκαμε με μεγάλη ταχύτητα, το εγκρίναμε όλα αυτά στις ε, εγκρίναμε τη γενική προσέγγιση στις 3 ε, Ιουνίου και συνεισφέρουμε με τρία μεγάλα βασικά στοιχεία. Είναι η διεύρυνση του όρου, της έννοιας του όρου για τη σωματεμπορίας, Επίσης, το θέμα της ποινικοποίηση των χρηστών ε, είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να γίνει γιατί δεν ισχύει στα κράτη, σε πολλά κράτη-μέλη μια τέτοια έννοια ε, και δύσκολα μπορεί να οριστεί το τι, ε, ε, ποιος θα έχει το βάρος της απόδειξης και ποιοι θα είναι αυτοί που θα πρέπει να τιμωρηθούν. Τώρα για τις ε, κυρώσεις, φυσικά και είναι σύμφωνο το Συμβούλιο, βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο θέλει να προχωρήσει πολύ περισσότερο. Επίσης, για το Συμβούλιο είναι πολύ σημαντικό η σημαντική προστασία που θα πρέπει να δίνεται στα θύματα για το θέμα των αδειών παραμονής ε, δεν είναι το Συμβούλιο που θα πρέπει να το εξετάσει. Θα υπάρξει ένα πρόβλημα νομικής βάσης φαντάζομαι. Η Κομισιόν πρέπει να το λύσει. Πρέπει να ακούσουμε τι θα μας πει. Όπως όμως και ο κύριος Δεκλέρκ το είπε χθε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η Βελγική Προεδρία εκφράζει την ικανοποίησή της που μπορεί να ξεκινήσει γρήγορα τις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει αυτό το μέσο να εγκριθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστώ. Για άλλα τρία λεπτά ο κύριος Μάικλ Κάρλιν, αν δεν κάνω λάθος, από την Επιτροπή. Ναι, ευχαριστώ πολύ. να ευχαριστήσουμε το Κοινοβούλιο για το σχέδιο έκθεσης που ευθυγραμμίζεται νομίζω με την πρότασή μας. Άρα το κείμενό σας πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το τελικό κείμενο. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα και σχόλια που έχουμε που κυρίως συνδέονται με το κατά πόσο αυτά τα θέματα θα έπρεπε να τα λύσουμε μέσω του νομοθετικού πλαισίου ή της στρατηγικής που σχεδιάζουμε για το 2011. Τώρα, πέντε θέματα που μας ανησυχούν, κυρίως τεχνικά, αλλά παρόλα αυτά μας ανησυχούν. Καταρχάς, πρώτη τροπολογία Νομική βάση το άρθρο 79. Να σας πω ότι αυτό μπορεί να περιπλέξει τη διαδικασία. Γνωρίζετε από τη συνθήκη ότι ορισμένες διατάξεις της θα έπρεπε να βασιστούν στο άρθρο 79 και άλλες στο 83. Έτσι θα καταλήγαμε σε ένα ευρυδικό σύστημα όσον αφορά τη νομική βάση, αν χρησιμοποιούσαμε το άρθρο 79. Και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα ερμηνείας και ενδεχομένως προβλήματα και με το δικαστήριο όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η νομική βάση γιατί θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Δεύτερον, κάποια πράγματα που αναφέρατε στην έκθεση. Για παράδειγμα, κατάσχεση των ε, παρανόμων εσόδων. Συμφωνούμε, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια του οριζόντιου πλαισίου για το οργανωμένο έγκλημα. Να υπάρξει δηλαδή μια νομοθετική πράξη γενικά για τις κατασχέσεις. Και έχουμε ξεκινήσει μελέτη αντικτύπου για αυτό το θέμα, άρα πρόκειται για προτεραιότητα για εμάς. Μετά, συντονιστής κατά της εμπορίας ανθρώπων. Είμαστε λίγο επιφυλακτικοί στο να αναφερθεί σε αυτό το έγγραφο Έχουμε δημοσιεύσει την προκήρυξη πριν από λίγες εβδομάδες και αύριο λίγη προθεσμία, οπότε θεωρούμε ότι θα έχουμε σύντομα τον συντηνιστή, αλλά παρόλα αυτά παραμένουμε επιφυλακτικοί στην αναφορά του εδώ στην πρόταση, καθώς αυτό το θέμα καλύπτεται από άλλη νομοθεσία. Τέλος, τροπολογία 45. Υπόδειξη ότι τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένα να καταστήσουν παράνομη τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Όπως είπε και το Βέλγιο, είναι λίγο δύσκολο το θέμα εδώ. Παρόλα αυτά θα θέλαμε να συζητηθεί το θέμα. Επί της αρχής λοιπόν επικροτούμε αυτή την πρόταση στην τροπολογία 45. Τέλος να πούμε ότι θα υπάρξει μία δήλωση όπου θα αναφερθούμε σε διάφορα σχετικά θέματα όσον αφορά την προσωρινή άδεια παραμονής. Η δήλωση θα γίνει το φθινόπωρο και τον Οκτώβριο θα κάνουμε μία εκτίμηση της κατάστασης όσο έχει σήμερα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ για τα σχόλια και σας ευχαριστώ γιατί ήσασταν συνοπτικός. Έχουμε 10 ομιλητές στον κατάλογο, παρακαλώ από δύο λεπτά ο καθένας. Ξεκινάμε τον κύριο Κίρκχοπ και μετά η κυρία Παρβάροβα. And I think that does make a slight difference to our contributions. I just want to say, first of all, that I understand that from a UK perspective, the current position of the government in the UK is to be opting out on this particular measure.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 Να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες γιατί έκαναν εξαιρετική δουλειά. Να υπογραμμίσω μερικά σημεία σύντομα. Και εγώ συμφωνώ να εγγυηθούμε την αρχή της μη απέλασης, δηλαδή να εγγυθούμε την παροχή άδειας παραμονής ε, στα θύματα. Διότι αλλιώς ε, και τα θύματα τα ε, βάζουμε στο ίδιο επίπεδο με τους θύτες. Και αυτό δεν είναι σωστό. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στην ομοθεσία κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων εγώ συμφωνώ ότι όποιος καταχράται ε, και εκμεταλλεύεται θύματα σωματεμπορίας θα πρέπει να διώκεται ποινικά. Σε περίπτωση τώρα ανηλίκων όλα αυτά διευρύνονται και συνδέονται άμεσα και με το σεξουαλικό τουρισμό που αντιμετωπίζεται στην οδηγία για την εκμετάλλευση των ανηλίκων. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ε, αναλύσουμε και να δούμε φυσικά την μελέτη επιπτώσεων της Κομισιόν. Η κυρία Έρνστ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν μεγάλες ευχαριστίες στους δύο εισηγητές που σε δύσκολα θέματα τα πήγαν καλά και δεν απέφυγαν δύσκολα θέματα έχουμε εδώ ε, αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Τώρα, κάποιε παρατηρήσει ε, που έχω, να τις συνοψίσω. Πρώτη παρατήρηση. Νομίζω και πάλι πρέπει να ξαναδούμε από το Α στο Ω όλα τα θέματα αυτή τη πρόταση και να εξετάσουμε κατά πόσον η πτυχή του φύλου λαμβάνεται επαρκώ. υπόψη. Υπενθυμίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι φυσικά, τα θύματα ε, ε, εμπορια ανθρώπων είναι γυναίκες τις περισσότερες φορές και πρέπει να δούμε κατά πόσον στα θέματα αυτά που εξετάζουμε και διατυπώνουμε αυτή η πτυχή του φύλου λαμβάνεται υπόψη και αντανακλάται. Δεύτερο σημείο, άτομα που πρέπει να προστατεύονται ιδιαίτερα. Παιδιά, για παράδειγμα, άτομα με μειονεξίες και άλλοι Πρέπει να προσθεθεί εδώ και η αμφίδρομη ε, ιδιότητα ε, δυνατότητας παραμονής. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό για να τους προστατέψουμε. Και επόμενο σημείο, πολλά αφορούν τον ορισμό εμπορία ανθρώπων. Αυτός ο όρος εμπορία ανθρώπων πρέπει να διαφοροποιείται και να διαφοροποιείται έναντι λαθρεμπορίας ανθρώπων. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε με σαφήνεια ποια πράγματα εντάσσονται σε αυτόν τον κύκλο εμπορίας ανθρώπων. Για παράδειγμα, την πρόσθετη μορφή της εκμετάλλευσης, παράδειγμα την ε, επαιτία, τη ζητιανιά. Θα πρέπει βέβαια εδώ να ε, διώκεται αυτή η πτυχή. Συμφωνώ με αυτό. Όμως από την άλλη πλευρά τη ζητιανιά δεν πρέπει να την ποινικοποιούμε ξεχωριστά. Πρέπει να προσέξουμε πολύ εδώ όποιος θέλει να το κάνει ας το κάνει. Αλλά όχι όμως ε, σε σχέση με τα παιδιά όταν είναι υποχρεωτική αυτή η δράση. Όμως υπάρχει και μια γραμμή διαχωριστική που δεν, μπορούμε να ξεπεράσουμε. Που έχει επιπτώσεις για παράδειγμα το ίδιο είπε και μια συνάδελφος ε, για την πορνεία πιο πριν. Το θέμα για την επαιτία, τη ζητιανιά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα παιδιά που για παράδειγμα τους ίδιους τους γονείς τους ας το πω έτσι, θα έπρεπε να, να θέσουμε υποδίωξη ποινική. Αυτά είναι θέματα περίπλοκα όσον αφορά τη ζητιανιά, την επαιτία για παιδιά και πρέπει να τα δούμε στη διατύπωσή μας. Επόμενο σημείο, πρόσβαση στη συνδρομή, νομική συνδρομή και συμβουλές. Πρέπει αυτή η νομική συνδρομή να είναι δωρεάν καταρχήν. Τελευταίο, τελευταίο σημείο, για τις αποζημιώσεις, επιτρέψτε μου να το πω, για την κατάσχεση και δίμευση είμαι υπέρ, αλλά πρέπει να σκεφτούμε αν μήπως κονδύλια Όροι για την επιβίωση αυτών των ανθρώπων, για τη διαβίωσή τους θα έπρεπε να διασφαλίζονται και να δίνονται σε αυτούς και θα, αυτό, αυτό θα πρέπει να το διατυπώσουμε. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που είμαι ομή και απότομη, αλλά γιατί διαφορετικά δεν θα λάβουν όλοι τον λόγο. Κυρία Σαζεντίνη, ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω πρόεδρε ως σκιώδης εισηγήτρια των Πρασίνων λαμβάνω τον λόγο. Θα ήθελα κάποια σημεία να αναφέρω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές πρώτα απ' όλα και επειδή αποφάσισαν από πλευρά τους ε, την ψυχή των ε, θυμάτων να την θέσουν στην ε, ανώτατη προτεραιότητα. Σε αυτή την οδηγία πρόκειται για πρόληψη λοιπόν. Έχουμε το θέμα της πρόληψης και πρόκειται επίσης και για καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων αλλά επίσης και για αντιμετώπιση της κατάστασης των θυμάτων και θέλω να πω ότι σε σχέση με την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων με διαφορετικού τρόπου μπορεί να διασφαλιστεί. Σίγουρα οι αυστηρότερε ποινέ ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα στην Ευρώπη, την μετανάστευση, διαδραματίζει και αυτό σε ένα ρόλο. Για να δώσω ένα παράδειγμα, προφανώ είναι ενδιαφέρον για κάποιου να απασχολούν παράνομου, επειδή είναι φθηνότερη η εργασία του και επειδή οι για παράδειγμα, σε θέσει εργασία εργασία στις επιχειρήσεις είναι ανεπαρκή. Εφόσον αυτό το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται θα έχουμε πάντα πρόβλημα. Άνθρωποι που είναι δηλαδή θύματα εμπορία ανθρώπων να οδηγούνται σε τέτοια κατάσταση. Και φυσικά θα μπορούσε κανεί να εξετάσει το θέμα της μη υποχρεωτική απέλασης όταν πρόκειται για θύματα. Όταν πρόκειται όμω για άδεια παραμονή που εξαρτάται από την δίκη έναντι ενό εμπόρου ανθρώπων, το, το πρόβλημα γίνεται, η κατάσταση γίνεται προβληματική. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Εξαρτάται πολλέ φορέ η διαδικασία από τέτοιε δίκε, από την έκβαση τέτοιων δικών, προτού μπορέσει να πάρει ένα τέτοιο άτομο άδεια παραμονή. Οι άλλοι που εκμεταλλεύονται τέτοιε υπηρεσίε ε, σίγουρα θα πρέπει ποινικά να διώκονται οι, εργαζο... οι εργοδότες τέτοιων παράνομων εργαζομένων διότι η ε, εκμετάλλευση τέτοιων υπηρεσιών είναι πολύ προβληματική υπόθεση Υπάρχουν διαφορετικέ απόψει στο Συμβούλιο και νομίζω και σωστά, διότι η ποινικοποίηση της παροχής υπηρεσιών στο τέλος, τέλο, τέλος πλήττει και ποινικοποιεί τα ίδια τα θέματα, της, τα θύματα με συγχωρείτε, της εμπορίας ανθρώπων. Και έτσι ε, τα δεινά τους συνεχίζονται και είναι πολύ πιο δύσκολο και να, ε, να δοθεί κάποια λύση. Τέλος, και διεξοδικά αναφέρθηκε αυτό και διακόπτει η Πρόεδρος. Παρακαλώ ολοκληρώστε. Βλέπετε κάποιο λόγο για να παρέμβετε. Ένα σημείο αν μπορώ να προσθέσω. Μερσή. Δύο λεπτά και διακόπτει η Πρόεδρος. Το τελευταίο μου σημείο αν επιτρέπετε Λοιπόν, διεξοδικά γίνεται αναφορά στο διαδίκτυο και σε μελέτες ε, και θα ήθελα να ε, ε, απευθύνω μια έκκληση. Τέτοιου είδους μέθοδοι δεν θα πρέπει να είναι απαντελώς ελεύθερες. Έχω υπόψη το εμπόριο ανθρώπων. Σας ευχαριστώ. Κώστια και μετά Διαστημέρα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για το εξαιρετικό της έργο και για τη συνεργασία που είχαμε για το γεγονός επίσης ότι λάβατε υπόψη σας διάφορα θέματα που πρότειναν οι σκιώδεις εισηγητής στην συνάντηση. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ξεκινάμε από ανθρωπιστική οπτική γωνία. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη σε όλα τα κράτη-μέλη και για τις κυρώσεις. Επίσης πρέπει να υπάρχει δωρεάν νομική βοήθεια. Αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν. Τρίτον, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των σημείων επαφής της Europol. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται για τους ανήλικους που είναι θύματα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως ίσως θα έπρεπε το Συμβούλιο να εξετάσει περισσότερο το θέμα και να δούμε πόσο ο Ευρωπαίος Συντονιστής θα μπορούσε να συνεργαστεί περισσότερο με την Europol, την Eurojust, το Frontex. Επίσης, να πω συμφωνώ με την τροπολογία 45, παρόλο που συνειδητοποιώ ότι θα δημιουργήσει προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη. Όμως σας υπενθυμίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά αυτά που προβλέπουν μια σειρά από κυρώσεις σε τέτοιε περιπτώσει. Τώρα όσον αφορά τη νομική βάση για την προσωρινή άδεια παραμονής. Όμως ίσως εδώ προκύπτει μια αντίφαση με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε περισσότερα τα θύματα και να τα ενσωματώσουμε στην κοινωνία. Όμως γνωρίζετε ότι το δικαίωμα παραμονής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από το αν θα γίνει προσφυγή από το θύμα και αν θα έχει επιτυχή έκβαση η δικαστική διαδικασία. Εκεί πρέπει να αλλάξουμε κάτι και στο ενδιάμεσο να δίνουμε αυτή την προσωρινή παραμονής. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε περισσότερο το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δίας Δεμέρα και μετά ο κύριος Φως. Εντάξει τώρα λειτουργεί, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στι εισηγήτρες ε, για μια τόσο σε βάθο δουλειά και τόσο περίπλοκη. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι αυτονόητο ότι όλη η προστασία πρέπει να διασφαλίζεται για τα θύματα. Οι επιφυλάξει, επιφυλάξει λακωνικότατα. Πρώτη επιφύλαξη. Λοιπόν, για το συντονιστή. Προσέξτε. Πρέπει να γνωρίζετε και φυσικά το γνωρίζει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουμε υπήρες ε, σύμβουλους, ε, ε, συνδέσμους ε, που ασχολούνται με αυτό το θέμα ακριβώς και πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό το Κοινοβούλιο και αυτή η, Ευρωπαϊκή, αυτή η Επιτροπή ε, εκπονούν μια έκθεση υπό συναπόφαση ώστε η συνέργεια και η αποτελεσματικότητα αυτής της διαμεσολάβησης να μπορεί να διαβιβάζεται στη Frontex. Είναι η, η ε, διασύνδεση με τις 27 ε, χώρες μέλη μέσω της Frontex. Και το επόμενο συμπίπτω με τους συναδέφους. Ο συντονιστής θα το συντονίζει όχι μόνο η Frontex αλλά η Ευρωπόλ και σε σχέση με την δίμευση και κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι ευρωβουλευτέ σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και με διαρμηνεί που είχαμε το προτέρημα να έχουμε την επαφή με Πασέα και μάλιστα και κλεισμένων των θυρών και σε ε, ε, αφρικανικέ ε, χώρε. Και υπάρχουν ακριβώ εδώ τα ίδια τα θύματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Κάποιοι τι κάνουν. Πρέπει να συμμερίζονται σε σχέση με τα θύματα αυτά την αγορά ε, και την, της βενζίνης για να κάνουν αυτή την ε, περατζάδα, αυτό το, αυτή τη διαδρομή. Και εδώ υπάρχει αυτή η μεταφορά των ε, αθών που περνάνε μέσω της, των Καναρίων νήσων στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι θύματα που φεύγουν από τη Σενεγάλη και πάνε στη, στα Κανάρια νησιά και δεν είναι οι Πακιστανοί. Η ποινικοποίηση των Χριστών. Αυτό βαίνει κατά του λόγου, του ορθού λόγου και της κοινή λογικής. Και για τα παιδιά. Τα παιδιά, πολύ σύντομα. Προσέξτε, για το Μάλι και την πολυγαμία. Έχουμε οικογένειες με 12 και 14 παιδιά. Αυτά τα παιδιά, επειδή δεν έχουν να φάνε, αφήνονται στις, ε, στα σχολεία και πρέπει εκεί να επιβιώσουν με κάποιο τρόπο. Ή έχουμε εδώ και ε, το θέμα αυτών των παιδιών, να το λάβουν υπόψη αυτό και στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Φως και μετά η κυρία Ρομέρο Λόπεθ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ως δικηγόρος θα ήθελα να αναφέρω πέντε πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινή πρακτική όσον αφορά την νομική ασφάλεια. Τροπολογίες 20 και 21. Εδώ έχουμε ποινές από 5 σε 6 χρόνια ή από 10 σε 12 χρόνια που αυξάνονται. Και θέλω να επισημάνω, αυτή η αύξηση δεν, δίνει δεν έχει αποτέλεσμα ε, αποτροπής. Βλέπουμε εδώ ότι διαρκώς υπάρχει δράση στο ποινικό τομέα και πολλές χώρες που ε, δεν μπορούν να πληγούν η συνεκτικότητα των νομικών των συστημάτων θα πρέπει να διασφαλιστεί στα κράτη-μέλη και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στα 5 και 10 χρόνια ως ποινές. Μετά, για το 22 βασανιστήρια και ψυχολογική βία. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι επαρκώ ακριβή. Έχουμε το κείμενο της 10 η Ιουνίου που είναι καλύτερο, είναι ακριβέστερο. Μετά για το 27 όταν ένα άτομο υπό καθεστώς βίας ε, ε, διαπράττει ένα ποινικό αδίκημα τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στη νομική ε, δίωξη και στην ποινή το γεγονό αυτό. Και στο άρθρο 7 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτό το θέμα. Το κείμενο του Συμβουλίου είναι καλύτερο. Εδώ τροπολογίες 29 και 30 στη συνέχεια. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ότι εδώ δεν είναι υποχρεωτική η ποινική δίωξη όταν κάποιο δεν, είναι, ε, δεν έχει την υπηκότητα του κράτου αυτού αλλά μόνο εθελοντικά μπορούν να δώσουν συνδρομή τα κράτη σε τέτοια περίπτωση γιατί αυτό θα οδηγούσε σε πολύ μεγάλες περιπλοκέ και προβλήματα και η τροπολογία 45 εδώ η επισήμανση σχετικά με αυτό ότι Πρόκειται για την ε, από πολιτικής πλευράς ε, η ελευθερία ε, κρίσης όσον αφορά την επιβαλόμενη ποινή λόγω του ότι η ποινή, οι πράξεις αυτές πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει ακριβώς ένα τέτοιο άτομο ότι έχει απέναντί του ένα τέτοιο άτομο και πρόκειται να διαπράξει ε, ποινικό αδίκημα. Και μετά η αποφυγή κατάθεσης, ε, αυτό θα περιέπλεκε τα πράγματα και θα τα επιβάρυνε αντί να τα διευκόλυνε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρωμέρο Λόπεθ και στη συνέχεια η κυρία Χίρς. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. θα ήθελα σε αυτά τα δύο λεπτά που έχω, μια και είναι ένα εγκάρσιο θέμα, οριζόντιο και αφορά πολλά θέματα, θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τη Σουηδική Προεδρία και ε, τι εισηγήτρες για τη δουλειά που έκαναν και θέλω να θέσω επιτραπέζη σε αυτό το θέμα που είναι σημαντικό για την πραγματικότητα στην οποία ζούμε σήμερα. Θα προσπαθήσω απλά και μόνο να εμείνω λίγο περισσότερο στην πτυχή των δικτύων, διότι είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιο είδος δικτύου όπως προηγούμενα αναφέρθηκε από ε, συνάδελφο. Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει με αυτό το πρόβλημα, με τα δίκτυα όσον αφορά το εμπόριο ναρκωτικών ή το εμπόριο ανθρώπων ή των μεταναστών, δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία και αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι μόνο το στα, τα, στατιστικά στοιχεία σημαντικό στοιχείο, αλλά και οι πληροφορίε για, το για αυτά τα φαινόμενα. Αν η Ευρωπόλ, για παράδειγμα, επιλαμβάνεται αυτού, δεν γνωρίζουμε μέχρι ποιού βαθμού έχουν δρομολογήσει επαρκείς μηχανισμούς για να αντιμετωπίζουν αυτά τα δίκτυα και να τα ξεριζώσουν. Διότι πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτού του είδους τα φαινόμενα αν δεν μπορούν να εκριζωθούν τελείως 100% τουλάχιστον να δουλέψουμε σε βάθος για να τα καταπολεμήσουμε. Είναι κρίμα ότι με αυτό το μέσο που έχουμε στα χέρια μας πρέπει να κάνουμε λόγο για δίμευση ή για αποζημίωση όταν είναι φαινόμενα αυτά τα οποία έχουν επιπτώσεις και στο οργανωμένο έγκλημα. Αλλά τέλος πάντων στην αναζήτηση αυτών των λύσεων καλό θα ήταν να επιμείνουμε σε κάποιες επιμέρους πτυχές ώστε εφόσον δεν έχουν συνολικά ληφθεί υπόψη σε άλλε οδηγίε, εδώ να καλύπτονται. Θα ήθελα να πω ότι εδώ θα έπρεπε να έχουμε και τον ανώτατο εκπρόσωπο τη Ευρωπόλ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα συγκεκριμένα και να ξέρουμε σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα τι υπάρχουν, τι στοιχεία υπάρχουν και για την καταπολέμηση τέτοιου είδου ε, δικτύων. Αν, έχουν, αν υπάρχει μια έκθεση από πλευρά του, μέχρι ποιο σημείο έχει επίπτωση αυτό σε σχέση με τι τρίτε χώρε από τι οποίε προέρχονται. Πρέπει να ξέρουμε την εμβέλεια του φαινομένου και το ε, ευρωπαϊκό ένταλμα ανακρίσεων και διερευνήσεων να μπορέσουμε να ε, το λάβουμε υπόψη γιατί έχει και αυτό τη σημασία του. Ευχαριστώ. Έχω δύο ακόμα αγορητές ε, στην, στον κατάλογο, όμως δεν έχουμε την Προεδρία ακόμα. Χίρς και μετά Μισελ παρακαλώ. Σε ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ως εισηγήτρια των φιλελευθέρων θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τις εισηγήτριες για αυτή την καλή συνεργασία. Να ευχαριστήσω επίσης για το γεγονός ότι η ιδέα μου της αποσαφήνισης ε, βρήκε α, απήχηση σε αυτή την εργασία. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτή την προσέγγιση. Η πτυχή, η συνιστόσα των θυμάτων να λαμβάνεται υπόψη, να ταυτοποιούνται πρώτα τα θύματα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να α, καταγράφονται, να αναφέρονται για τις επαγγελματικές ομάδες που συσχετίζονται να υπάρξει ευαισθησία γιατί μπορεί να πρόκειται ακριβώς για τέτοιου είδους θύματα ανθρώπινης εμπορίας. Είναι σημαντικό σημείο αυτό και είμαι ευγνώμων για την τροπολογία 14 όπου στοχευμένα η κατάρτιση και η εκπαίδευση τέτοιων ατόμων προβλέπεται που έχουν σχέση με τέτοια άτομα στην Γερμανία για παράδειγμα ε, το γεγονός της εμπορίας ανθρώπων δεν χρησιμοποιείται πολλές φορές στη Γερμανία υπάρχουν πολλές φορές αβεβαιότητες ε, ανασφάλειες και εδώ σε σχέση με το αξίωμα του συντονιστή θα ήθελα σύντομα το αναφέρω αν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ένα αξίωμα ένα, μια θέση όπως συντονιστού εργασίας ή ε, δραστηριοτήτων θα πρέπει να προαχθεί αυτό. Και θα ήθελα να προσθέσω τη φωνή μου στις προλαλήσασες για την τροπολογία 45, για την κατηγορία των ε, όσων εκμεταλλεύονται τέτοιες ε, δυνατότητες. Έχουμε και το πρόβλημα της απόδειξης ε, στοιχείων. Πώς αποδεικνύουμε ότι κάποιος γνώριζε ότι είχε απέναντί του ένα θύμα εμπορίας ανθρώπων. Και το άλλο θέμα είναι, και δεν πιστεύω ότι αυτό είναι υπέρ της πρόληψης, όταν εκ των υστέρων βλέπει κάποιος ότι έχει απέναντί του ένα θύμα Εμπορία ανθρώπων, τότε αυτό το άτομο δύο φορές θα το ξανασκεφτεί αν ο ίδιος ή το ίδιο αυτό άτομο θα ε, διακυβεύσει την ασφάλειά του σε σχέση με παραβάσεις που έχουν ε, ε, γίνει όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων με το άτομο αυτό. Χαίρομαι για το ότι μπορούμε να εργαστούμε προς αυτόν τον κοινό στόχο και όλα αυτά θα μπορέσουν να ευδοκιμήσουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος, ο κύριος Λουί Μισερ και μετά σύντομα θα επανέλθουμε στις εισηγήτριες. Ο κύριος Μισελ. Πάρα πολύ σύντομα κυρία μου. Εγώ θα επανέλθω στο, στην τροπολογία 45 όπου αναφέρεται για τους κινδύνους που βαρύνουν ε, τους ε, χρήστες ε, κυρίως όταν πρόκειται για στρατιωτικούς λόγους κλπ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω καθόλου, μα καθόλου δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτή η προσθήκη. Εγώ συμφωνώ αρκετά με την συνάδελφο για να πούμε ότι το θέμα της πορνείας δεν μπορεί να λυθεί από αυτήν την οδηγία. Εγώ θα ήμουν υπέρ να έχουμε μία ειδική οδηγία για την καταπολέμηση της πορνείας. Είναι κάτι το πολύ πιο πολύπλοκο, το πολύ πιο δύσκολο, πιο σύνθετο για να το βάλουμε εδώ. Θα έπρεπε λοιπόν να πάμε σε μία διαφορετική οδηγία. Συγχαίρω πάνω στις εισηγήτριες για την εξαιρετική τους εργασία. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σύντομος. Οι συγητές παρακαλώ πολύ γρήγορα γιατί έχουμε εδώ τον Υπουργό. Πολύ σύντομα. Εμένα μου φάνηκε να κατάλαβα ότι η τροπολογία 45 ε, ε, ερμηνεύθηκε διαφορετικά στις διάφορες γλώσσες Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό το 45. Στην ε, μετάφραση ε, έχει γίνει μία παρανόηση. Δεν ποινικοποιούμε τις υπηρεσίες, αλλά αυτούς που καταχρώνται των θυμάτων συνείδητα. Ξέρω ότι ορισμένοι συνάδελφοι έχουν πρόβλημα σχετικά με το βάρος της απόδειξης. Θα κοιτάξουμε να βρούμε τη λύση. Η πορνεία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως αποκλειστικό θέμα αυτής της έκθεσης γιατί θα υπάρξουν αμφισημίες μπορούμε να εξετάσουμε και την πορνεία γιατί το 4% των θυμάτων της σωματεμπορίας καταλήγουν στην πορνεία. Το θέμα όμως της έκθεσης δεν είναι αυτό. Διευκρίνηση λοιπόν για την τροπολογία 45 θα γίνει σύντομα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπάουερ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Τρία σύντομα σχόλια. Όσον αφορά τον ορισμό, υπάρχει Ευρωπαϊκή Σύμβαση, υπάρχει το, Παλέρμο του πρωτο, το πρωτόκολλο του Παλέρμου, με συγχωρείτε, όπου επίσης υπάρχει πολύ συγκεκριμένος ορισμός. Τώρα, όσον αφορά τα άτομα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πολλές περιπτώσεις ε, όπου έρχονται τα θύματα από την Αλβανία, από τη Σερβία, από τρίτες χώρες δηλαδή, αλλά που έχουν άδεια παραμονής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήταν λάθος να διώκονται. Όσον αφορά τώρα την τροπολογία 45, ο βασικός λόγος δεν ήταν να τιμωρηθούν όσοι έλαβαν μεταμόσχευση και εκ των, προτέρων, εκ των υστέρων προέκυψε ότι το όργανο προέρχονταν από θύμα εμπορίας. Καταλαβαίνουμε ότι κινδυνεύει η ζωή τους. Όμως υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου γίνεται σκόπιμα η διαδικασία και αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Επίσης, όσον αφορά τη σχέση πορνείας και εμπορίας, είναι διακριτά θέματα. Σε κάποιες χώρες είναι παράνομη η πορνεία, σε κάποιες άλλες όχι. Γι' αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το θέμα της πορνείας και να επικεντρωθούμε στα θύματα εμπορίας. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτησή μας. Ευχαριστώ την συμπρόεδρο, την κυρία Σφένσον. Θα Ζητήσω τώρα από τον Υπουργό, τον κύριο Βατλέ, να κάτσει δίπλα μου. Σας ευχαριστώ που υπομείνατε και την συζήτησή μας λίγο γιατί καθυστερήσαμε. Συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Αν θέλετε να συζητήσετε, παρακαλώ, εκτός εθούσης. θα ήθελα να υποδεχθώ εκ μέρους της Επιτροπής Δημόσιων Ελευθεριών των... κύριο Μπατλέ που είναι Υπουργό ε, της ε, Βελγικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τη μετανάστευση και την πολιτική ασύλου, την πολιτική για την οικογένεια. Μακρύς ο τίτλος. Γνωρίζουμε όλοι ότι η πολιτική ασύλου είναι στην ημερήσια διάταξη ως προτεραιότητα. Τους επόμενους έξι μήνες θα συζητηθούν κάποια σημαντικά θέματα. Σας δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Προεδρίας. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω για την ε, υποδοχή στην Επιτροπή σας και να θυμίσω πόσο Σημαντική είναι η πολιτική μετανάστευσης και ασύλου είναι μια πολιτική ιδιαίτερα σημαντική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Είναι πραγματικά λοιπόν πολύ σημαντικό στην αρχή της προεδρίας, μιας προεδρίας να δίνουμε τις γενικές γραμμές που θα ακολουθήσει η Βελγική Προεδρία στην, κατά τη διάρκεια της. Επίσης, η Βελγική Προεδρία εντάσσεται στη γενική ε, γραμμή συνέχειας ε, των προηγουμένων ε, προεδριών για την μετανάστευση και το άσυλο υπάρχουν ήδη σημαντικά έγγραφα υπάρχει και η συνθήκη της Λισαβόνας δηλαδή έχουμε ένα σωρό νομικά κείμενα τα οποία πλαισιώνουν την πολιτική στην οποία θέλει να εγγραφεί και το Βέλγιο ως Προεδρία και για αυτό το θέμα και για πολλά άλλα το Κοινοβούλιο μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας έχει επιπλέον εξουσίες και το Κοινοβούλιο πλέον είναι ο σημαντικός πρωταγωνιστής ε, για τα θέματα αυτά με τις ευαισθησίες του, με τα μηνύματα που θέλει να στείλει και που θα πρέπει να ενσωματώσουμε στα νομικά μας κείμενα και στις εφαρμοστικές πολιτικές αυτών των κειμένων για τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Επίσης ε, θέλω να θυμίσω ε, να σας ε, πω μάλλον ήδη εισαγωγικά ότι είμαι έτοιμος να έχουμε όλες ε, τις συζητήσεις που χρειάζονται για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Πρέπει να έχουμε έναν κοινό στόχο και ο στόχος μας πρέπει να είναι μια κοινή πολιτική ασύλου για το 2012 και για να γίνει πραγματικότητα κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε την στενή συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ποια είναι τα μεγάλα θέματα που θέλουμε να εξετάσουμε κατά την Προεδρία. Τέσσερα. Πρώτον, εναρμόνιση για το άσυλο. Δύο, διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης. Τρία, καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Και τέσσερα, πολιτική ενσωμάτωση. Όλα αυτά καταδεικνύουν σε ποιο βαθμό εμείς θέλουμε να διαμορφώσουμε μια ισορροπημένη πολιτική μετανάστευσης και ασύλου που θα εγγράφεται ε, ως ε, άθροισμα όλων αυτών των πολιτικών. Θέλουμε να έχουμε και πολιτικές για την νόμιμη μετανάστευση αλλά και την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Θέλουμε όμως να έχουμε και πολιτική ενσωμάτωσης. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αποτελούν τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση για το άσυλο. Ο στόχος ε, για το κοινό καθεστώς ασύλου το 2012. Έχουμε έξι νομοθετικά κείμενα τα οποία εκκρεμούν σχετικά. Και ξέρουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ συγκεκριμένα στα πλαίσια της Βελγικής Προεδρίας για ορισμένα από αυτά. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέσα σε αυτήν την προοπτική δηλαδή του κοινού πακέτου. για τις οδηγίες Eurodac, δηλαδή των μακράς διαρκείας ε, διαμενόντων, και για το Δουβλίνο μπορούμε να προχωρήσουμε για να ξεκινήσουμε αυτό το, για να κατακτήσουμε μάλλον αυτό το πρώτο βήμα για μια κοινή πολιτική το 2012. Έχουμε και τα δύο κείμενα που αφορούν στην διαδικασία και την οδηγία για την υποδοχή είναι κείμενα τα οποία δεν είναι τόσο προχωρημένα ως προς την πολιτική συνένεση αλλά είναι εξίσου σημαντικά και θα πρέπει να τα προχωρήσουμε και αυτά. Βέβαια δεν φαντάζομαι ότι κατά την Προεδρία μας θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την έγκριση των δύο και αυτών κειμένων που σας ανέφερα. Θα συνεχίσουμε όμως να εργαζόμαστε. Διότι έχουμε ορισμένες οριζόντιες διαστάσεις ιδιαίτερα σημαντικές Θα μπορέσουμε λοιπόν με όλη αυτή την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα τέσσερα πρώτα κείμενα που θα αποτελέσουν και το πρώτο στάδιο του συνολικού πακέτου για την ολοκλήρωση δηλαδή του στόχου ε, για, το, για την κοινή πολιτική ασύλου το 2012. Δεύτερο έχουμε την νόμιμη μετανάστευση. Γνωρίζουμε ότι το κείμενο για την ενιαία άδεια είναι ένα κείμενο που συζητήθηκε, συζητιέται. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν θα έρθει με προτάσεις για τους εποχιακούς εργαζόμενους και θα μπορέσουμε κατά τη Βελγική Προεδρία να εξετάσουμε αυτά τα τρία κείμενα. με τις ε, τους, δηλαδή για τους εποχιακούς εργαζόμενους και τους εργαζόμενους ICT. Δεσμεύτηκε, είπαμε, η Κομισιόν να έρθει το Σεπτέμβριο με προτάσεις. Για το άσυλο και την μετανάστευση, πέρα από αυτό το κοινό καθεστώς ε, για το άσυλο και την νόμιμη μετανάστευση, Έχουμε φυσικά και τη συνέχιση της πολιτικής για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Το Frontex θα πρέπει να ξανασυζητηθεί, πρέπει να προχωρήσουμε. Ανακλείσω το τηλέφωνο μου, λέει ο Προεδρεύων. Μαθαίνω πάντα. Λοιπόν, για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης πρέπει να δούμε με, τι θα κάνουμε με τα θέματα επανεισδοχής, με όλες αυτές τις διαδικασίες που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα για τη Βελγική Προεδρία είναι το θέμα των μη συνοδευομένων ανηλίκων. Γνωρίζετε ότι στο τέλος της Ισπανικής Προεδρίας παρουσίασε ένα κείμενο η Κομισιόν, το συζητήσαμε στο Συμβούλιο. Στα πλαίσια της Βελγικής Προεδρίας θα οργανώσουμε μία διάσκεψη για αυτό το σημαντικό θέμα των μη συνοδευομένων. Ξέρω ότι είναι μία πολύ δύσκολη και σημαντική προβληματική. Θέλουμε να ανταλλάξουμε τις καλές πρακτικές, να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη για τους μη συνοδευομένους ανηλίκους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης και του ασύλου. Αυτό έχει να κάνει με τη συνεργασία μας ε, ε, και τις σχέσεις μας για θέματα μετανάστευσης με τις Ηνωμένε Πολιτείε και τη Ρωσία, όπως επίσης και το θέμα που, ε, τις γενικές συζητήσεις που έχουμε για το θέμα των θεωρήσεων και την απολευθέρωση των θεωρήσεων θα το προσέξει ιδιαίτερα το θέμα το Βέλγιο, κυρίως στον τοσχέ που αφορά στη Βοσνία και στην Αλβανία, όπου γνωρίζετε ότι έχουν σταλεί εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε τα συμπεράσματά τους για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προχωράμε στα πλαίσια αυτών των προβληματικών. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Εμείς ε, το ξέρουμε ε, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και για αυτά τα θέματα. Και για να τελειώνω και να αφήσω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στις ερωτήσεις και στην ανταλλαγή απόψεων, ε, να σας πω ότι το δικό μας όραμα για αυτήν την Προεδρία είναι κυρίως να ακούσουμε τα μηνύματα που μας έχει στείλει το Κοινοβούλιο να πετύχουμε την πιο ισορροπημένη πολιτική μετανάστευσης και ασύλου εν ώψη του 2012 και να προχωρήσουμε επίσης και στα θέματα νόμιμης μετανάστευσης και να έχουμε μία προσέγγιση όσο το δυνατόν πιο αλληλέγγυα μεταξύ των κρατών μελών. Πρόκειται για τη συζήτηση σε επίπεδο Δουβλίνου αλλά και η γενική εναρμόνιση για θέματα ασύλου. Επίσης καταπολέμηση της λάθρομετανάστευσης προχωρώντας στον τοσχέ του Frontex αλλά και τα θέματα ενσωμάτωσης ε, που πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι φιλόδοξοι στόχοι. Ανταποκρίνονται. Πιστεύω και στις επιθυμίες του Κοινοβουλίου για θέματα μετανάστευσης είναι όμως ταυτόχρονα και ένα ισορροπημένο πρόγραμμα για να μπορέσει να δώσει ακριβώς αυτή την προπτική μας, αυτή την προπτική που θέλουμε για την ολοκλήρωση σε θέματα μετανάστευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Έχω κάποιους ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο Προτείνω να ξεκινήσουμε με δύο-τρεις ερωτήσεις μαζί, να απαντήσετε και μετά να ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Δίας Νεμέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υφυπουργέ. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας και άκουσα σε το τέταρτο σημείο να μιλάτε για ολοκλήρωση, για ενσωμάτωση, συγγνώμη. Δεν το αναφέρατε βέβαια το θέμα, δεν το αναπτύξατε γιατί ακριβώς η ενσωμάτωση των μεταναστών δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Εγώ απαγοητεύτηκα λίγο με αυτά που μας είπατε για το πακέτο ε, του ασύλου. Ε, είχαμε πει να ολοκληρώνουμε το 2010, δεν το βλέπω όμως. Ε, εντάξει, συμφωνώ, έχουμε την Eurodac, έχουμε το Δουβλίνο, αλλά με απαγοητεύει αυτό το θέμα. Και κάτι άλλο που με ανησυχεί. Θέλω να ξέρω σε τι συνίστανται όλες αυτές οι αποστολές μετανάστευσης σε τρίτες ε, ε, χώρες. Θέλω να ξέρω τι σημαίνει αυτό που έχουμε στο βελγικό πρόγραμμα. Διότι φαντάζομαι ότι έτσι θα έχουμε και, και, επικάλυψη αρμοδιοτήτων ε, με τους υπαλλήλου της ΕΙΣΕ, τις οποίους έχουμε. Ήδη είναι καμιά τριανταριά δηλαδή και αυτοί όλοι οι σύνδεσμοι, οι υπάλληλοι σύνδεσμοι που έχουμε αποσπασμένους ε, εργάζονται για τα θέματα του Frontex. Ε, λοιπόν, ε, τελευταίο κύριε Υφυπουργέ, θέλω να ξέρω για τον κανονισμό Frontex. Τι θα κάνει συγκεκριμένα η Βελγική Προεδρία, τι νέες αρμοδιότητες θα, θα ενταχθούν στον κανονισμό Frontex. Η κυρία, Ρομέρο και μετά Βίγκστρομ και μετά θα απαντήσει ο Υπουργό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Πάλι θα περιορίσω το χρόνο ομιλίας γιατί έχουμε πάνω από 10 άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο και χρειαζόμαστε και χρόνο για τις απαντήσεις του Υπουργού. Παρακαλώ λοιπόν σύντομα. Ευχαριστώ για τις ε, εξηγήσει που μα έδωσε η Βελγική Προεδρία για όλα αυτά τα θέματα. Θέλω να ρωτήσω, καταρχήν, ο κύριος Λετέρμα μίλησε για κατάχρηση του ασύλου, του δικαιώματος ασύλου κατά την παρουσίαση του προγράμματος της Βελγικής Προεδρίας. Τι νόημα έδωσε ο κύριος Λετέαγμα σε αυτόν τον όρο κατάχρηση. και ορισμένες χώρες μπορεί να θεωρούν ότι γίνεται κατάχρηση του ασύλου αλλά εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι και πολύ περήφανη για την ομοθεσία της σχετικά. Θέλω να ξέρω τι νόημα έδωσε ο κύριος Λετέγμα σε αυτό και όσον αφορά στο φύλλο πορείας ε, και την εφαρμογή του για τις διαδικασίες τίθενται όλα αυτά ως προτεραιότητα στην πολιτική ασύλου. Ποια είναι λοιπόν τα οριζόντια εμπόδια στην ολοκλήρωση της ε, οδηγίας για τις διαδικασίες. Επίσης, για την κοινή πολιτική μετανάστευση υπήρχε μια, ένα κοινό σύμφωνο, μια συμφωνία κοινή για τη μετανάστευση η οποία τελικά σε τι χρησιμεύει μόνο στην οργάνωση κοινών πτήσεων για επαναπατρισμό. Έχετε προβλέψει λοιπόν να προχωρήσει κάτι, έχετε κάποιες πρωτοβουλίες σχετικά. Ευχαριστώ κυρία Βέξτρομ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την εισήγηση που έγινε από πλευράς Υφυπουργού. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και θέλω να πω ότι συμπίπτουμε στι απόψει και εύχομαι κάθε επιτυχία στη Βελγική Προεδρία σε συνεργασία με εμά, με την Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή. Όσον αφορά την Eurodata, και όσον αφορά την μακρά διάρκεια άδεια παραμονή, υπάρχουν δυνατότητε να μπορέσουμε να στοχεύσουμε στην σωστή νομοθεσία. Δύο οδηγίε είναι πολύ σημαντικέ. Η υποδοχή Reception και η Procedure Directive, η οδηγία διαδικασιών. Ανησυχώ κάπως ότι αυτά μπορεί να οδηγήσουν να αγνοηθούν κάποια πράγματα προσπαθώντας να στοχεύσουμε σε μια τέτοια ρύθμιση. Πρέπει να προσέξουμε, είναι δύο πολύ σημαντικές οδηγίες. Αν αφαιθούν κάποια πράγματα εκτός, τότε θα διακυβευθούν πράγματα για το μέλλον που δεν θα μπορέσουν να ρυθμιστούν σωστά και έτσι θα αλλάξουμε και την έννοια όλα ε, της ε, ε, φιλανθρωπίας ή της ανθρωπιάς και γι' αυτό είναι σημαντικό αυτές τις πτυχές να τις λάβουμε υπόψη. Παρακαλώ λοιπόν αυτό τον κίνδυνο να τον αντιμετωπίσετε με σοβαρότητα. Να θεσπίσετε ένα χρονοδιάγραμμα πότε εμείς ως Κοινοβούλιο μπορούμε να αναμένουμε από εσάς ότι η οδηγία για την υποδοχή θα μπορέσει να ευδοκιμήσει. Εκείνο που θέλουμε είναι πραγματικά να γνωρίζουμε πότε θα δοθεί συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία. Και πρόκειται και για μια έκκληση αλλά και για μια παράκληση. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Ευχαριστώ. Κύριε Βακλέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ για αυτές τις πρώτες ερωτήσεις. Να απαντήσω στον κύριο Δίας Δεμέρα, το πρόφερα σωστά το όνομά σας μάλιστα. Εγώ μίλησα για το κεφάλαιο ενσωμάτωση. είναι πολύ σημαντική αυτή η πολιτική. Είναι σίγουρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άμεσες αρμοδιότητες σχετικά, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες κοινέ δράσεις και θα πρέπει να αναπτυχθούν. Δεν μπορούμε εμεί να, βλέπουμε, να αντιμετωπίζουμε την πολιτική ασύλου και μετανάστευση χωρί να εξετάζουμε και αυτό το κεφάλαιο γιατί δεν θα, μας δεν θα μπορέσουμε αλλιώ να προχωρήσουμε εύρυθμα. Για το Frontex πρέπει να του δώσουμε τα ίδια μέσα, τα ίδια μέσα να έχει δηλαδή το Frontex να πρικοδοτηθεί και με κονδύλια και προσωπικό για να προχωρήσει. Υπάρχει, είπαμε, το στοιχείο για της παράνομης μετανάστευσης και το στοιχείο της ολοκλήρωσης και υπάρχουν και τα στοιχεία που ανέφεραν η κυρία Ρομέρο και η κυρία Βόλστρομ σχετικά με την οδηγία για τις διαδικασίες που αναφέρατε και οι δύο που είναι επίσης πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να προχωρήσουμε σχετικά έχοντας πάντοτε ως στόχο την κοινή πολιτική ασύλου για το 2012. Εσείς μας είπατε ναι, είχαμε πει πρώτα 2010. Ε, λοιπόν, 2012 είναι τώρα, δεν πρέπει να χάνουμε λοιπόν χρόνο. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το πρώτο βήμα. Eurodac, ανταλλαγή ε, η πληροφόρηση, Δουβλίνο είναι ε, η πολιτική ε, που εξισορροπεί και τα θέματα αρμοδιοτήτων και ευθυνών με την αλληλεγγύη. Υπάρχει η εναρμόνιση Έχουμε λοιπόν επίσης και το θέμα των καλυφικασιών, δηλαδή των όρων ε, για, την, ε, για τον προσδιορισμό. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να εξεταστούν κατά την ε, Βελγική Προεδρία. Και αυτά εν ώψη του ορίζοντα του 2012. Κυρία Ρομέρο Λόπες αναφέρατε και το λόγο του Πρωθυπουργού μας, του κυρίου Λετέρν. Το Βέλγιο φέτος με την απολευθέρωση των θεωρήσεων αντιμετώπισε τεράστιες ροές ζήτησης βίζας από τις ε, χώρες με τις οποίες έγινε το άνοιγμα. Και αυτό λειτουργήσε εις βάρος των όσων ζήτησαν τη βίζα τελικά που είχαν λάθος ενημέρωση. Δηλαδή ήρθε εδώ ένα σωρό, κόσμος ο οποίος νόμιζε ότι παίρνοντας τη θεώρηση ε, για το Βέλγιο, ερχόμενο στο Βέλγιο θα είχε διασφαλισμένη εργασία, στέγη, τροφή. Γι' αυτό λοιπόν πριν προχωρήσουμε στη χορήγηση θεωρήσεων θα πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο των χωρών που θα τη χάνουν ελεύθερης θεώρησης. Πρέπει λοιπόν να τους ενημερώνουμε ούτως ώστε να μην πέφτουν θύματα λανθασμένων πληροφοριών από διάφορους εκμεταλλευτές που τους λένε «Λάτε στο Βέλγιο θα έχετε κοινωνική ασφάλιση, δουλειά κλπ. Χρειάζεται λοιπόν ένα monitoring για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία απολευθέρωσης των θεωρήσεων. Και όσο περισσότερο έχουμε μια καλύτερη εξέλιξη ε, <coughs> στην απολευθέρωση των θεωρήσεων, τόσο πιο καλά θα λειτουργήσουν τα πράγματα και στις οποίες ε, δίνονται ελεύθερες ε, θεωρήσεις και για τους κατοίκους τους. Συνεχίζουμε με Αργεντίνη Ταβάρες Κλάς από δύο λεπτά ο καθένας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ουάτλε, κύριε Υπουργέ, το κείμενο της Βελγικής Προεδρίας το είδα όσον αφορά το άσυλο και την μετανάστευση. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου Τώρα, αν θα το καταφέρουμε να πετύχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου με κάτι τέτοιο, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Αυτό που θέλετε να πετύχετε μέχρι το Δεκέμβριο, <clears throat> δηλαδή για μια τροποποίηση σε σχέση με το Δουβλίνο, καλό θα ήταν, διότι αναμένει το Κοινοβούλιο μια τέτοια δράση και όχι μόνο το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχουν Αυγανοί, για παράδειγμα, που αποστέλλονται στην Ελλάδα και εκείνοι αναμένουν. Και διαβάζω επίσης την πρότασή σας τοποθετήσεις της Βελγικής Προεδρίας για συμφωνίες λέει με τρίτες χώρες. Γίνεται λόγος εδώ για τη Λιβύη. Μια Ευρωπαϊκή Αφρικανική Σύνοδος Κορυφής θα διεξαχθεί λέει το, τον, ε, το φθινόπωρο. Και εδώ πρέπει να δούμε την επίγευση με βάση αυτά που συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα. 400 υπηκόσεις της Ερυθρέας που προσπάθησαν να καταλήξουν στην Ιταλία τους ε, επέστρεψαν οι Λίβοι πίσω προς την χώρα τους. Θα έλεγα λοιπόν, αν και όταν η Ευρώπη κάνει λόγο για μετανάστευση και άσυλο, πρέπει να γίνει λόγος για την προστασία των ανθρώπων που έχουν δικαίωμα για να τύχουν ασύλου. Και το σημαντικό είναι μια καλή πολιτική μεταναστευτική πολιτική γιατί είναι υπεργυρασμένη η κοινωνία μας και χρειαζόμαστε τους μετανάστες. Βλέπω ότι είναι γενικόλογες οι τοποθετήσεις στο κείμενό σας. Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το τι θα πρέπει να γίνει και να επιτευχθεί. συμφωνούμε μέχρι το Δεκέμβριο 2010 να υπάρξουν προτάσεις, να αναμείνουμε λοιπόν και να δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος ε, Ταβάρες μετά Κλάς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και σε σχέση με τις ε, παρεμβάσεις από πλευράς ε, της ομάδας μας που θα υπάρξει και παρεμβάσει από τον συνάδελφο, εγώ θα περιοριστώ στους ε, μετανάστες και την επανεγκατάσταση, που είναι και τα θέματα μου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στις εκθέσεις που έχω προετοιμάσει και που δεν βρίσκω ανάμεσα στις προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας κάτι σε σχέση με αυτά. Λοιπόν, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτά τα σημεία σε αυτά τα θέματα. Εργαζόμαστε τους τελευταίους μήνες για αυτά τα θέματα, τα, ζητήματα αυτά με μεγάλη συνένεση στην Ευρωβουλή. Οι δύο εκθέσεις ε, που εγκρίθηκαν τον προηγούμενο Μάιο με την έγκριση 500 ψήφων μεγάλη συνένεση και έχουμε συγκεκριμένες ιδέες για την μονάδα επανεγκατάστασης ε, ή την πολιτική επανεγκατάστασης ε, μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της ε, ΕΑΣ. Και υπάρχουν επίσης και κάποια εγκάσια οριζόντια θέματα πολύ σημαντικά για τις delegated actions, τις κατεντολήν, κατεκτέλεση αρμοδιότητες ανάληψης δράσης και θα πρέπει να μπορέσουμε να εργαστούμε για αυτά γιατί είναι ζητήματα τα οποία αναφύονται και με διάφορες εκθέσεις. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό θέμα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει ακριβώς αυτά τα οποία θα έπρεπε. 5.000 πρόσφυγες ετήσια επανεγκαθιστούμε. Όταν 80.000 επανεγκαθιστούν είπα, οι συνολικές ανάγκες είναι 200.000 ε, για 200.000 πρόσφυγες ετήσια και αν κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας, αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να επιληθεί σε ε, παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτή την πτυχή και ελπίζω να δω περισσότερα από την Βελγική Προεδρία για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. τελευταίο σε αυτό το γύρο, κύριος Κλάς. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη για το κινητό, το μικροφωνισμό. Κύριε Γουατλέ, πρέπει πραγματικά να πω ότι είναι... μας να ακούμε ότι η Βελγική Προεδρία την παράνομη μετανάστευση, λέει, θα καταπολεμήσει. Λέω με έκπληξη το αναφέρουμε, διότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική της βελγικής κυβέρνησης είχε τέτοια μορφή, ώστε η παράνομη μετανάστευση προαγόταν αντί να καταπολεμάται. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο συλλογικό πρόβλημα τη ενόησης των παράνομων μεταναστών νομιμοποίησής τους ε, που 10 20 χιλιάδες για παράδειγμα επιμέρους χατοφυλάκια νομιμοποίησης εκκρεμούν. Μυριάδες λοιπόν παράνομοι αλλοδαποί υπάρχουν υφίστανται στο Βέλγιο που ανταμείβονται με άδεια διαμονής και αυτό αντιβαίνει σε αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει η Ευρώπη και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών μέσα στη ζώνη της, ε, της ζώνης Σέγγεν για ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Ερώτησή μου, ποια συγκεκριμένα μέτρα προβλέπετε λοιπόν, τι θα προτείνετε στο Συμβούλιο για την καταπολέμηση της ε, παράνομης μετανάστευσης, διότι όταν βλέπω την κατάσταση στο Βέλγιο είναι διαφορετική. Και όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση, κάνετε λόγο για μια κύρια προτεραιότητά σας, λέει, για αυτό το θέμα. Θέλετε την μετανάστευση νέων μέτρων, την υιοθέτηση νέων μέτρων να λάβετε υπόψη για την προαγωγή της νόμιμης μετανάστευσης για να καταπολεμηθεί η υπεργύρανση στην Ευρώπη. Και εξετάζεται, λέει, την ε, μετανάστευση εργαζομένων προς την Ευρώπη ή δημογραφικής ανανέωσης. Έχουμε εκατομμύρια άνεργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως σήμερα. Τι θα γίνει με όλους αυτούς όταν εσείς λέτε ότι η αγορά εργασίας θα επωφεληθεί από την νόμιμη μετανάστευση. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος να απολεστούν από το σύστημα αυτά τα άτομα που είναι άνεργα σήμερα. Και όταν είσαστε υπέρ μιας ενιαίας διαδικασίας, λες και μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να επιλύσει όλα τα προβλήματα, πώς μπορούμε να αποφύγουμε να καταλήξουν σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά τα άτομα όπου δεν θα υπάρχει εργασία για ε, Ευχαριστώ. Καταρχάς για την κυρία Σαργεντίνη σας ευχαριστώ γιατί αυτό που μας ζητάτε είναι να προχωρήσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα και να προχωρήσουμε σε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να προχωρήσουν αυτά τα νομοθετικά κείμενα. Βεβαίως, έχω σαφώς προτεραιότητες. Το αναφέρουμε και στο πρόγραμμα της Προεδρίας. Υπάρχουν τέσσερα θέματα και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι πιο σαφής όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και του σαφείς στόχους της Βελγικής Προεδρίας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ταβάρας ε, για το ερώτημα. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα του επαναπατρισμού. Είστε και εισηγητής προκύπτουν πολλά ερωτήματα συχνά θα δούμε και τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν. Υπάρχει θέση του Βελγίου και έχει συμμετέχει το Βέλγιο στη διαδικασία αυτή του resettlement, της ε, επανεγκατάστασης. Πρόκειται για ένα θέμα που είναι σημαντικό και ενδιαφέρει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο ερώτημα του κύριου Κλάς να σας υπενθυμίσω ότι στο Frontex είναι από τους πιο δραστήριους εταίρους ε, το Βέλγιο, το ίδιο και όσον αφορά τη μετανάστευση. Άρα αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας ε, και βεβαίως ε, με βάση και τη μελλοντική δημογραφική πρόκληση για την Ευρώπη πρέπει το Βέλγιο και οι χώρες μας όλες να αντιμετωπίσουν αυτές τις ε, προκλήσεις τις δημοκρατικές στο μέλλον και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσει η Ευρώπη στο μέλλον. Σας ενημερώνω αγαπητοί συνάδελφοι ότι έχουν ζητήσει άλλοι 8 το λόγο. Κλείνω εδώ την λίστα των ομιλητών και αν όλοι παραμείνετε όσο σύντομοι ήταν οι προλαλήσαντες θα καταφέρουμε να τελειώσουμε στις 11. Για κουλίνο παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Καλωσορίζω τον προεδρεύοντα, ο οποίος μίλησε για υπευθυνότητα, αλληλεγγύη, έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και όλα αυτά φυσικά εγγράφονται στο έγγραφο της Στοκχόλμης βάσει του οποίου θα θέλαμε εμείς οι ευρωπαϊκές αρχές να συμβαδίσουν. Αναφέρατε δύο οδηγίες για τους εποχιακούς εργαζόμενους από τρίτες χώρες και την μεταφορά τους στις επιχειρήσεις που τους απασχολούν. Και όλα αυτά βεβαίως συνδεδεμένα και με τη γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Πιστεύετε ότι κατά το ευρωπαϊκό ε, βελγικό εξάμεινο θα το λύσετε το πρόβλημα και χάνετε το μικρόφωνο του ομιλητή. Σε τι συνίσταται για, τους, τη Βελγική Προεδρία η αλληλεγγύη. Όλες οι παράλληλες χώρες αντιστέκονται με νύχια και με δόντια στην παράνομη μετανάστευση και προσπαθούν και συνάπτουν διμερείς συμφωνίες. Μα πότε η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει να συνάπτει αυτές τις συμφωνίες. Δεν είναι πρόβλημα αυτά της ε, Ελλάδας, Ιταλίας, της Μάλτας, της Κύπρου. Όλα αυτά δεν είναι ε, ε, παρεστήσεις ορισμένων από μας είναι πραγματικές ανάγκες που απαιτούν να περάσουμε σε ένα στενότερο σύστημα συνεργασίας, ένα ευρωπαϊκό σύστημα συνεργασίας. Η κυρία Γκυγιόμ, ευχαριστώ. Εσείς φαντάζομαι θα καταλάβατε για το άσυλο πόσο σημαντικό είναι για μας από τις ερωτήσεις που σας έγιναν και θα κάνω κι εγώ επίσης μια ερώτηση καταλάβαμε ότι θέλει η προεδρία να ολοκληρώνει το συντομότερο δυνατόν ορισμένα κείμενα αλλά αν ορισμένα από αυτά τα κείμενα περάσουν και εγκριθούν να ξέρετε ότι άλλα δεν θα περάσουν δεν θα προχωρήσουν και δεν θα καταλήξουν πουθενά. Οπότε αν υπάρξει μία απόλυξη για το άσυλο τελικά θα έχουμε κάτι το εντελώς ανισόρροπο διότι θα πρόκειται για κάτι το οποίο θα, έχει, ε, θα απορρέει όχι από τα βασικά κείμενα αλλά από παράγωγα κείμενα Θα πρόκειται λοιπόν για κάτι το εντελώς ετερόκλητο και θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη που είχαμε και στην πρώτη φάση επεξεργασίας του κειμένου. Επίσης ε, η πραγματικότητα πολλές ε, φορές ε, μπορεί να είναι πολύ πιο σκληρή στην πραγματικότητα. Ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη επιμένουν ιδιαίτερα στο θέμα του κόστους όλων των ε, μέτρων που αφορούν στο άσυλο. Εγώ κατάλαβα ότι έχετε ένα χρονοδιάγραμμα της Προεδρίας για πολλά κείμενα αλλά υπάρχει και ένα θέμα οριζόντιο που έθεσαν ορισμένοι συνάδελφοι. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες δουλειές που έχει ολοκληρώσει η Κομισιόν για τα οριζόντα λύσεις. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και δεν έχουμε αντίστοιχες ε, πραγματικότητες για τις διάφορες θεματικές. Θα μπορούσαν ε, λοιπόν να αποτελέσουν τη βάση για να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε, αλλά εγώ θα σταματήσω τώρα. Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Είμαι υπεύθυνο για το Frontex και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου μέχρι το τέλος του έτους. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πού βρισκόμαστε όσον αφορά το φάκελο Frontex στο Συμβούλιο και συγκεκριμένα πού βρισκόμαστε στην ε, πιθανότητα να αγοράσει δικό του εξοπλισμό το Frontex ε, τα πλαίσια του οράματος ε, για μετατροπή του σε ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή. Δεύτερον, μετά από αυτά που είπε και ο κύριος ε, Ιακολίνο για την ε, αλληλεγγύη, θα ήθελα να πω ότι η πολιτική μετανασύλου βασίζεται στην αλληλεγγύη αλλά θα θέλαμε να δούμε αλληλεγγύη όχι μόνο για τους σε άσυλο αλλά και για τις ε, χώρες που αντιμετωπίζουν δυσανάλογα μεγάλες πιέσεις. Δεν αναφέρεται τίποτα στο κείμενό σας για αυτές τις χώρες και αυτή την αλληλεγγύη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι σκοπεύει να κάνει η Βελγική Προεδρία για αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ίσως θα μπορούσα να απαντήσω στο ερώτημα των κυρίων Διακολίνο και Μπουσουτήλα για την αλληλεγγύη. Θεωρώ ότι το Δουβλίνο είναι μια διαδικασία που μας ε, επιτρέπει να κάνουμε κάτι κατά αυτόν τον τρόπο, να διαπιστώσουμε πότε βρίσκεται υποπίεση ένα κράτος μέλλον και αυτή την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί. Γνωρίζετε κύριε Μπουσουτήλο ότι υπάρχουν για παράδειγμα διατάξεις όσον αφορά την επανεγκατάσταση όπου περιλαμβάνονται διατάξεις αλληλεγγύης. Υπάρχει επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο, υπάρχει ο μηχανισμός υποστήριξης ε, σε επίπεδο Frontex. Υπάρχουν λοιπόν πρακτικά μέτρα που σας βοηθούν και βεβαίως πρέπει να περάσουμε σε καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Πάντως, αυτή η αλληλεγγύη πρέπει να ιδωθεί παράλληλα με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη εναρμόνιση για το σύστημα ασύλου προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα μηχανισμό αλληλεγγύης που θα έχει νόημα όταν οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο όραμα. Πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε τη συζήτηση για την αλληλεγγύη με τη συζήτηση για την υπευθυνότητα όντως υπάρχουν χώρες που αντιμετωπίζουν τεράστιες πιέσεις και πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη προς αυτές. Παράλληλα όμως πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη εναρμόνιση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών και έτσι αυτό το όραμα που έχουμε για το άσυλο θα προβλέπει πολύ μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος, αυτό το μείγμα που δεν είναι καθόλου εύκολο να επιτευχθεί πολιτικά. Αλληλεγγύη και υπευθυνότητα. Τώρα, για το Frontex. Να πω ότι ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες προόδους όσον αφορά το Frontex Χρειαζόμαστε τους ε, ίδιους πόρους και άλλα πράγματα προκειμένου να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του Frontex και πιστεύω ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στην ε, συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο ερώτημα της κυρίας Γκυγιό για την πρώτη φάση, αν θέλετε. Μας ενδιαφέρουν κυρίως οι, οι υποχρεώσεις στο θέμα του qualification, του προσδιορισμού. Έχουμε ένα κείμενο που δεν είναι απολύτως αυτόνομο. Προσπαθούμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μια στάση όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένη, όπου σε πρώτη φάση έχουμε και την πτυχή Eurodac και την πτυχή αλληλεγγύη και υπευθυνότητα στα πλαίσια του Δουβλίνου και την πτυχή επιμακρών διαμενόντων και προσδιορισμός τους. Όπως είπα λοιπόν και προηγουμένως, πρέπει πάντα να προχωρούμε με στόχο το να επιτύχουμε πρόοδους. Παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις βρισκόμαστε μακρύτερα από μία συμφωνία από ό,τι σε άλλες. Όμως αυτή η κοινή προσέγγιση μπορεί να μας οδηγήσει στην επιτυχία των στόχων μας για το 2012. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να παραμείνει αυτή η πρώτη φάση που μου φαίνεται απαραίτητη. Και περνάω στο τελευταίο ερώτημα για την νόμιμα μετανάστευση του κυρίου Γιακολίνη. Έχουμε το πακέτο που αφορά τους εποχικούς εργαζόμενους στα ICT και τους μόνιμους και αυτό το πακέτο θα το μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Σε ένα γύρο όλοι οι υπόλοιποι ομιλητές. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τον Υφυπουργό μου φάνηκε να κατάλαβα ότι μας διασφαλίσατε την βαθιά στράτευση της Βελγικής Προεδρίας ως προς τον καταμερισμό των ευθυνών των κρατών μελών αλλά και τον καταμερισμό των υποχρεώσεων σχετικά με την ενσωμάτωση. Εμείς ε, θέλουμε να δούμε και απτά στοιχεία αυτής της βούλησης. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας ε, να ε, προχωρήσετε πιο γρήγορα το ντοσιέ για τους μη συνοδευομένους ανηλίκους ε, που είναι προτεραιότητα της Βελγικής Προεδρίας. Τελευταία ερώτηση τώρα. Συζητήσαμε μόλις την πρόταση οδηγίας για την σωματεμπορία και τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι να ισχύει η μη απέλαση για τα θύματα της σωματεμπορίας να δίνουμε δηλαδή άδεια παραμονή σε αυτούς που έχουν, είναι βεβαιωμένα θύματα ε, της σωματεμπορίας. Θέλω να ξέρω ποια είναι η απάντησή σας, η κυρία Χιμένες. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό και θα ήθελα να του πω ότι έρχομαι από την Ισπανία και πιο συγκεκριμένα από την, Ανδαλουσία. Εμείς εκεί υποφέρουμε ιδιαίτερα από τη λαθρομετανάστευση. Στο Μοτρίλ κοντά στην Γρανάδα πρόσφατα βούλιαξε μια σχεδία όπου πνίγηκαν και δυο μωρά ε, δηλαδή και όπου εμείς πάμε διακοπές και κάνουμε τα μπάνια μας ε, λοιπόν, ε, εσείς ε, είπατε ότι χρειάζεται πληροφόρηση, πληροφόρηση για τις χώρες οι οποίες υπόκεινται το μεγαλύτερο βάρος. Μα νομίζω ότι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Κάθε μέρα γράφεται στις εφημερίδες. Θα παρακαλούσα λοιπόν τη Βελγική Προεδρία να κοιτάξει η αλληλεγγύη μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών να γίνει πραγματικότητα. ούτως ώστε οι χώρες του Νότου να μην αντιμετωπίζουν μονάχες τους το πρόβλημα της υποδοχής. Εγώ, να εμένα μου στέλνουν γράμματα από, χωριουδάκια στην, ε, ε, και μου λένε τι προβλήματα έχουνε και ο κύριος Γιακολίνο το είπε. Λοιπόν, πραγματικά μην το ξεχάσετε αυτό το πρόβλημα. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι δεν είμαι σίγουρη πραγματικά ότι απαντήθηκαν πολλές ερωτήσεις από αυτές που διατυπώθηκαν και που ήταν ενδιαφέροντα τα θέματα τους. Θα προσπαθήσω λοιπόν πολύ εξειδικευμένες ερωτήσεις να κάνω και καλό θα ήταν να παίρναμε και εξειδικευμένες απαντήσεις αν γίνεται. Πρώτα απ' όλα για την Frontex. Δεν θέλω να ξέρω η Βελγική Προεδρία στοχεύει να ξεκινήσει διακριβωτικές έρευνες για τις φήμες και τις τοποθετήσεις ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με ρεφουλμό των ατόμων που συλλαμβάνονται. Θα υπάρξει ανάκριση, αν όχι γιατί. Και θα ήθελα επίσης να επιμείνω στην ερώτηση του κυρίου Μπούσουτιλ. Ποια είναι η δική σας άποψη, η άποψη της Βελγικής Προεδρίας. Πού θα έπρεπε να ενταχθεί η Frontex, τι θα έπρεπε να γίνει σε πέντε χρόνια με τη Frontex, πώς θα πρέπει να μετεξελιχθεί και πώς θα διασφαλιστεί το δικαίωμα σε άσυλο με όλα αυτά σε σχέση με ένα άλλο θέμα. Υπήρξε κάποια αντίσταση από ό,τι γνωρίζω στο Συμβούλιο κατά μια κοινή πολιτική για το άσυλο. Μεταξύ άλλων και από τη Γερμανία η αντίσταση αυτή. Πώ στοχεύετε να ξεπεράσετε αυτέ τι αντιστάσει, τι θα κάνετε και πότε σχεδιάζετε να ξεπεραστούν τα προβλήματα ώστε να κινητοποιηθούμε προ τα εμπρό, προ μια κοινή πολιτική ασύλου. Και ποια είναι η στρατηγική σα για τι προτεραιότητε για την νόμιμη μετανάστευση. Και τελευταία ερώτηση, πώ σχεδιάζετε να κινηθείτε στο μέλλον όσον αφορά την Ελλάδα που δεν έχει ένα πραγματικό σύστημα ασύλου. Τι θα κάνει η Βελγική Προεδρία για την περίπτωση της Ελλάδας ώστε να είναι ασφαλεί οι πρόσφυγες εκεί και να μπορούν να ετούνται άσυλο στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Πολλέ ερωτήσεις που έχουν στριμωχτεί σε λιγότερο από δύο λεπτά. Κυρία Έρνστ παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα, ο εναρμονισμός του δικαιώματος, του δικαίου για το άσυλο είναι πολύ σημαντική υπόθεση και η προλαλή σας θα το ανέφερε ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από τη Γερμανία και γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας ποια είναι. Τι θα κάνετε ώστε αυτές οι επιφυλάξεις της Γερμανίας να, να ξεπεραστούν, να τις αντιμετωπίσουμε κάπως. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής. Πρώτη, εσείς στο πρόγραμμά σα διατυπώσατε ω Βελγική Προεδρία και είπατε ότι το επίπεδο ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται. Υψηλό επίπεδο ασφάλεια για του ετούντε άσυλο. Όταν πρόκειται για εναρμονισμό του ε, δικαίου περί το άσυλο. Διατυπώνεται ότι πρέπει αυτοί που πρέπει να την χάνουν προστασία να προστατεύονται. Ποιου έχετε υπόψη πρώτον όσον αφορά τον τομέα του ασύλου ώστε να επεκταθεί αυτό το δικαίωμα. Ποια ε, διατύπωση θα χρησιμοποιηθεί. Το δεύτερον, γίνεται λόγο για μια αποτελεσματική σύμφωνη συμφωνία επαν, και επιστροφής και νέες συμφωνίες λέει θα, δια, θα συναυθούν με άλλες χώρες. Τι θα ξεκινήσει και πώς ξεκινά η Προεδρία σας σε αυτό τον τομέα. Τρίτον, όσον αφορά συνόδευτα ανήλικα παιδιά, μη συνοδευόμενα ανήλικα παιδιά που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Τι θα γίνει συγκεκριμένα, εξειδικευμένα για αυτά τα παιδιά. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Πραγματικά τα μη συνοδευόμενα παιδιά, τα ανήλικα, να προστατεύονται ιδιαίτερα. Να υπάρχει δυνατότητα λήψη απόφαση ε, για αυτά. Τι θα γίνει. Υπό το πρίσμα ότι πιθανόν θα έχουν την ευκαιρία να παραμένουν, να παραμείνουν στη χώρα τους υπό συγκεκριμένε ε, προϋποθέσεις. Ζητήθηκε και για την Frontex να τοποθετηθείτε. Αδημονώ να ακούσω ποιες είναι οι απόψεις σας για την Frontex, ε, πράγμα το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση τώρα. Ευχαριστώ. Τελευταία κυρία Φαγιόν παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες. Πολύ σύντομα, στο Κοινοβούλιο είμαι υπεύθυνη για την φιλελευθερωποίηση των θεωρήσεων για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και θα ήθελα να σας ζητήσω περισσότερες συγκεκριμένες πληροφορίες ε, για το θέμα γιατί είπατε ότι είναι προτεραιότητα της Βελγικής Προεδρίας. Όμως ε, είμαι λίγο αποτυγοητευμένη από τη συμπεριφορά της Βελγικής Προεδρίας ε, γιατί δεν βλέπω το Βέλγιο να προσπαθεί ιδιαίτερα να καταλήξει κάπου με τις δύο αυτές χώρες οι πληροφορίες μου λένε ότι οι χώρες αυτές είναι τεχνικώς έτοιμες, αλλά στο τελευταίο πρόγραμμα της ε, Βελγικής Προεδρίας αναφέρεται ότι οι Υπουργοί θα συζητήσουν το θέμα τον Νοέμβριο και όχι τον Οκτώβριο όπως είχε προγραμματιστεί. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ε, υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης ή κάτι άλλο. Να σας πω επίσης ότι το προηγούμενο Νοέμβριο μαζί με το Συμβούλιο είχαμε καταλήξει σε μία κοινή δήλωση. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο, αλλά εσείς από ό,τι φαίνεται όχι. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Δύο μιλητές αναφέρθηκαν στη σωματεμπορία. Το Βέλγιο τον Οκτώβριο έχει προβλέψει μία διάσκεψη σχετικά για να απαντήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης σχετικά με την σωματεμπορία. Ευχαριστώ τις κυρίες Έρνστ και Αντζελίλη που τόνισαν το θέμα των μη συνοδευομένων ανηλίκων. Είναι θεμελιώδες το ζήτημα. Μπορούμε να μιλήσουμε για την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ κρατών μελών για των μη συνοδευομένων ανηλίκων πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτήν την ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα που είναι οι μη συνεδευόμενοι ανήλικοι. Για την κυρία Χιμένες, μα φυσικά εμείς έχουμε συνειδητοποίηση ποια είναι η πίεση που δέχονται οι εκτεθειμένες στη μετανάστευση χώρες. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε αυτήν την πολιτική που θα συνδέει την ευθύνη με την αλληλεγγύη για το Frontex. Το είπα πριν και στον κύριο ε, Μπουσουτήλ. Χρειάζονται, χρειάζεται να προχωρήσει. Ε, ευχαριστώ και την κυρία Κέλλερ που ξανά ε, είπε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα εναρμονισμένο σύστημα για το άσυλο. Είναι ουσιαστικότατο Πρέπει λοιπόν να παίξουμε το ρόλο μας και να παίξει και το Κοινοβούλιο το ρόλο του. Άκουσα από πολλούς ε, τη βούληση ε, να προχωρήσουμε εν ώψη του 2012. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Πρέπει όμως ε, να προχωρήσουμε για την καλύτερη εναρμόνιση για το θέμα της κυρίας Έρνστε σχετικά με το υψηλό επίπεδο προστασίας Όλοι έχουμε υπογράψει τη σύμβαση της Γενέβης και όλοι πρέπει να κάνουμε, ε, να προχωρήσουμε στην αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα για να μπορέσουμε να καταστήσουμε σεβαστή την σύμβαση της Γενέβης όσο το δυνατόν πιο εναρμονισμένα στην επικράτειά μας. Θα πρέπει επίσης να επιμείνουμε ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε από από κοντά όλες τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει και με το Μαρόκο και με την Τουρκία και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στις συμφωνίες επανεισδοχής είναι ένα μέσο σημαντικότατο για την άσκηση πολιτικής ασύλου χρειάζεται, είναι δύσκολο να επιτευχθούν όλες αυτές οι συμφωνίες αλλά τον επαναπατρίστε κάποιον χωρίς να έχετε άδεια επανεισδοχής είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό βλέπω ότι συζητάτε σήμερα, το, ψηφίζετε σήμερα το θέμα της επανεισδοχής με το Πακιστάν. Τώρα για την απολευθέρωση των θεωρήσεων. Δύσκολα να σας εκφράσω την άποψή μου πριν να έχω την έκθεση ε, των εμπειρογνωμόνων που έστειλε η Κομισιόν στην Βοσνία και στην Αλβανία. Πρέπει να δούμε πώς οι χώρες αυτές πληρούν τους όρους που τους έχουν επιβληθεί. Και η ανάλυση πρέπει να γίνει με όσο το δυνατόν περισσότερη αντικειμενικότητα. Θα σας πούμε περισσότερα στοιχεία όταν μας απαντήσουν οι επιρρογνώμονες Κομισιόν. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Νομίζω ότι υπάρχουν ένα-δύο ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Αν έχετε χρόνο, θα ήθελα να σας ζητήσω να ακούσετε και αυτές τις ερωτήσεις και μετά να απαντήσετε γραπτός. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις που ήδη έχετε κάνει στη Γραμματεία για να τις αποστείλουμε γραπτό στον Υπουργό και να λάβουμε γραπτή απάντηση. Μόνο τις ερωτήσεις που είχατε κάνει τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ψηφοφορία για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πακιστάν για την επανεισδοχή. Ο κύριος Σόγκορ είναι ο εισηγητής. Σας υπενθυμίζω ότι χρειάζεστε την κάρτα ψηφοφορίας σας. Βάλτε την παρακαλώ στη σχισμή. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Μία αιτιολόγηση, επεξήγηση ψήφου της πολιτικής μας ομάδας. Μετά πολλές διαπραγματεύσεις και συζητήσεις μεταξύ μας αλλά και με την Επιτροπή και συγκεκριμένα την κυρία Μάλστρομ, η ομάδα μας θα ψηφίσει υπέρ γιατί λάβαμε μία εγγύηση και μία δέσμευση. Λάβαμε μία γραπτή εγγύηση όπου υπενθυμίζεται σαφώς από την Επιτροπή η διεθνής προστασία και η υποχρέωση μη επαναπατρισμού που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αν υπάρχει σαφής πιθανότητα σημαντικών βλαβών για το άτομο αυτό στην χώρα καταγωγής του. Λάβαμε λοιπόν σημαντικές δεσμεύσεις από την Κομισιόν επίσης για να πιέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρησιμοποιώ τον όρο ακριβώς που χρησιμοποίησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επικυρώσει το Πακιστάν ε, τη σύμβαση της Γενέβης και Κάθε έξι μήνες θα ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Κοινοβούλιο για την εφαρμογή των συμφωνιών επανιστοχής. Αυτό θα ισχύει και για το Πακιστάν καθώς και για τα αποτελέσματα των Μικτών επιτροπών. Και επίσης ε, δημιουργία ενεργών επαφών με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Άρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει μια πολιτική ευθύνη να δράσει και να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις της. Αυτό θα κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι δεσμεύσεις μας δεν αφορούν μόνο τις χώρες, αφορούν και το Κοινοβούλιο από πλευράς Επιτροπής έχετε όλοι μπροστά σας αυτή τη γραπτή δέσμευση της Επιτροπής και γι' αυτό το λόγο θα ψηφίσει υπέρ η ομάδα μας. Ευχαριστώ κυρία Γκρινσπεκ. Τρία ακόμη άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν είναι συζήτηση, αλλά κάποιοι θέλουν να κάνουν σχόλια επί της ψηφοφορίας. Κυρία Φλότρ, παρακαλώ. όντως ε, μια επεξήγηση ψήφου μπορεί να γίνει μετά τη ψηφοφορία αλλά αφού ξεκίνησαν ε, τώρα να μιλήσω και εγώ χωρίς ε, να θέλω να δυσκολέψω την προεδρία σας. Θα ήθελα λοιπόν να επιβεβαιώσω ότι μετά από πολλή σκέψη οι πράσινοι δεν θα συμφωνήσουν με αυτή τη συμφωνία επανεσδοχής με το Πακιστάν γιατί πρόκειται για την πρώτη χώρα υποδοχής προσφύγων στον κόσμο και τα συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται δεν μας δείχνουν ότι η δέσμευση της Επιτρόπου για την εφαρμογή Επιτόπου θέματα που έχουν να κάνουν με τα ταξιδιωτικά έγγραφα όταν δεν υπάρχει λεσεπάσε και τα λοιπά Εκεί υπάρχουν προβλήματα παρά και τις διαβεβαιώσεις του πρέσβη του Πακιστάν, οπότε εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτή την πρώτη συμφωνία επανεισδοχής που εξετάζεται στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας. Ναι κύριε Πουσουτήλ, σας έχω δει. Οι υπόλοιπε επεξηγήσει ψήφου μπορούν παρακαλώ να είναι πολύ σύντομε. Ένα λεπτό παρακαλώ. Επί διαδικαστικού, κύριε Μπουσουτήλ. Αυτή η διαδικασία είναι σε καμία περίπτωση μάλλον δεν είναι σύνομη με την διαδικασία. Παρακαλώ ξεκινήστε αμέσως τη ψηφοφορία. Ορισμένα μέλη ήρθαν εδώ μόνο για την ψηφοφορία. Δεν προβλέπεται χρόνος για συζήτηση, μόνο για ψηφοφορία. Όταν ζητάει κάποιο το λόγο δεν μπορώ να γνωρίζω εκ των προτέρων τι πρόκειται να πει. Κύριε Κέρκοπ, έχετε ζητήσει διαδικαστικό. Μετά θα κάνουμε την ψηφοφορία και μετά θα περάσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Ναι, συμφωνώ κυρία Πρόεδρε. Και σύμφωνα με τον κανονισμό, οι επεξηγήσεις ψήφου γίνονται πάντα μετά την ψηφοφορία, όχι πριν. Πριν γίνεται μόνο η συζήτηση επί του θέματος Νομίζω ότι υπάρχει άρθρο του κανονισμού που αναφέρει ότι πρώτα έχουμε την ψηφοφορία και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που θα το τηρήσετε. Ευχαριστώ. Τώρα η ψηφοφορία μετά σύντομες επεξηγήσεις. Παρακαλώ, περνάμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζετε υπέρ αν συμφωνείτε με τη συμφωνία, διαφορετικά κατά η αποχή. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινάει τώρα. Ψήφισαν όλοι. Όχι. Παρακαλώ αλλάξτε μηχάνημα. Κυρία Γιαρόκα, μπορείτε να αλλάξετε θέση. Δούλεψε. Τελειώσαμε. Ένα άτομο δεν έχει ψηφίσει ακόμη. Πέρας ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται 30 υπέρ 22 κατά καμία αποχή. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής έχει ζητήσει το λόγο. Πρώτα λοιπόν παίρνετε εσείς το λόγο και μετά περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Κύριο Σόγκορ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπεψήφισαν. Oh, Συγγνώμη, δεν υπήρξε λέει διερμηνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω απλά του συναδέλφους για τη σοφία τους όσους υπεψήφισαν. Ευχαριστώ. Η πιο σύντομη παρέμβαση που έχουμε ακούσει. Παρακαλώ, όσοι φεύγετε ήσυχα. Η κυρία Ένστ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να ε, δηλώσω και να ε, κάνω και μια τοποθέτηση. Εμείς ως GUNGL Ενωτική Αριστερά, Βόρεια Πράσινη Αριστερά, καταψηφίσαμε αυτή τη συμφωνία. Επειδή έχει ρόλο κλειδιού για μελλοντικέ συμβάσει και συμφωνίες. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε και στις άλλες περιπτώσεις μελλοντικά και σε αυτήν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πολιτικά δικαιώματα δεν διαδραματίζουν κάποιο ρόλο. Βλέπουμε τώρα ότι δεν μας ικανοποιούν οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοσμητικού χαρακτήρα εξοραίζουν τα πράγματα και δεν είναι επί της ουσίας. Και έχουμε μεγάλη ανησυχία όσον αφορά τους πρόσφυγες για ε, πολλά θέματα. Φοβόμαστε ότι δεν θα υπάρξει κατάλληλη προστασία των προσφύγων. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση της Γενέβης το Πακιστάν, άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα προστατεύσουν επαρκώς τους πρόσφυγες. Θα συμφωνήσω λοιπόν με άλλους συναδέλφους και με την Ελέν Φλότρ και θα καταθέσουμε μία έκθεση μειοψηφία που θα στείλουμε σε όλους τους συναδέλφους ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συνυπογράψουν. Κυρία Γκυγιόμ, πολύ σύντομα είχαμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε τη θέση μας ως πολιτική ομάδα. Είχαμε θέσει πολλά ερωτήματα και λίγες ε, σαφείς απαντήσεις λάβαμε. Όσον αφορά τις ε, δεσμεύσεις εντός εισαγωγικών της Κομισιόν δεν είναι αρκετή πρόοδος και να πω ότι αυτές τις δεσμεύσεις εντός εισαγωγικών Τις είδαμε και χτες πώς η Επιτροπή ασχολείται με τα θέματα επανιστοχής και τις συμφωνίες. Ελπίζουμε πάντως ότι όντως θα λαμβάνουμε ενημέρωση κάθε έξι μήνες για τις νέες συμφωνίες και να πω ότι και εμείς θα έχουμε έκθεση μειοψηφίας. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε εδώ αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στο σημείο 11 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Δύο θέματα παρουσίαση των επιπτώσεων της συνθήκης της Λισαβόνας και ενδεχομένως ε, συζήτηση με εκπρόσωπο της μόνιμης Επιτροπής για την Εσωτερική Ασφάλεια, της Επιτροπής Κόζη. Δεν ξέρω ακόμη αν έχει επαληθευτεί αυτό. Πάντως, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει αύξηση των ευρωπαϊκών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρέπει να βρεθεί ένα γενικό πλαίσιο που θα καλύπτει την ενισχυμένη συνεργασία αυτών των οργανισμών αλλά και των οργανισμών με τα εθνικά και ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Επίσης ε, πρέπει να ασχοληθούμε με την μόνιμη Επιτροπή για την Εσωτερική Ασφάλεια καθώς και γενικά το σχεδιασμό της Επιτροπής για την Πολιτική Ασφαλείας. Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης σκοπεύει η Κομισιόν να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, ειδικά όσον αφορά τις ε, τους οργανισμούς όπως η Europol και η Eurojust που πρόκειται να ενταχθούν στη Λισαβόνα. Αν όλα αυτά δεν γίνουν εγκαίρως θα καθυστερήσουμε αρκετά. Είχαμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την ε, που θα ξεκινήσει με την ε, Jean Lambert. Μετά πρέπει να ε, παληθεύσουμε αν έχουμε κοντά μας τον κύριο Κούκομπερτ. Ναι, τον έχουμε. Ωραία, η κυρία Λάμπερτ τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου εκπρόσωπο της ΛΥΜΕ διότι στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα που υπάρχει στην διακομματική θεσμική ομάδα για τις, ε, ε, ε τους οργανισμούς και υπηρεσίες ε, συναποτελείται από εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Είμαι όμως σε σχέση με αυτά τα θέματα η μόνη που έχει για παράδειγμα επαφές με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Το παρασκήνιο είναι ο έλεγχος του προϋπολογισμού που πρέπει να πούμε ότι ε, η εξέταση του έργου των υπηρεσιών με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνεται. Λοιπόν, το θέμα είναι τι γίνεται σε σχέση με τη συμφωνία, με την συνθήκη της Λισαβόνας και την ημερήσια διάταξη της Λισαβόνας και σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η γραμμή του Κοινοβουλίου καθορίζεται από την έκθεση Παπαστάμκου του 2008. Έχουμε εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και εκπροσώπους ε, της ε, γραμματείας με συγκεκριμένα συγκεκριμένους, ε, συγκεκριμένες επαφές σε οργανισμούς ε, και υπηρεσίες. Και η ΛΥΜΠΕ, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, συνδέεται και προσπάθεια είναι να βρούμε κοινέ προσεγγίσεις όσον αφορά την διοργάνωση και την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιών και οργανισμών και να δούμε αν μπορούν κοινέ αρχές να ισχύουν και να θεσπιστούν για τη δομή τους, για τη λειτουργία τους και τον έλεγχό τους. Από την άλλη πλευρά υπάρχει πολυμορφία μεταξύ των οργανισμών όπως βλέπουμε και ένα από τους τομείς που συζητούμε είναι σίγουρα ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πραγματικά, με άλλα λόγια, πώς ένα από τα θέματα δηλαδή που θα εξετάσουμε κάποια στιγμή είναι και πάλι ένα το οποίο θέτει το Κοινοβούλιο για τη δομή και τον διάλογο και τη διαβούλευση των οργανώσεων και υπηρεσιών με τους εμπλεκόμενους που διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό. Να έχουμε δηλαδή μια πλήρη εμβέλεια αξιολόγησης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλους τους οργανισμούς και υπηρεσίες που και για όσους ενδιαφέρονται για ένα θερινό ανάγνωσμα στην παραλία θα το συνιστούσα γιατί λίμπε υπάρχει ένα, ε, ας το πω έτσι, υπάρχουν δεδομένα που μπορούν να διοχετευτούν και να διανεμηθούν από τη γραμματεία. Όμως κάποια θέματα έχουν μεγαλύτερη σημασία. Κάποια από αυτά ως αντίδραση από πλευράς μας στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Θα πω δύο λόγια σε σχέση με αυτό και για το ψήφισμα του Νοεμβρίου 2009. Όπως είπατε, Πρόεδρε, δύο υπηρεσίες, κυρίως η Eurojust και η Europol, τώρα έχουν καθεστώς, ας το πω έτσι, συνθήκης αναγνωρίζονται στα άρθρα 85 και 88 σε, συνθήκη, σε, επίπεδο συνθήκης και επίσης και για τη θέση των Εθνικών Κοινοβουλίων εξίσου όσον αφορά την αξιολόγηση υπό το εθνικό πρίσμα για τις δραστηριότητες των οργανισμών και υπηρεσιών και επίση για αυτή τη συγκεκριμένη Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όχι μόνη τη αποκλειστικά, αλλά υπάρχουν θέματα για τι συμφωνίε και συνεργασία με τρίτες χώρε, που είναι κάτι το οποίο γνωρίζω ότι απασχόλησε την Κοινοβουλευτική αυτή Επιτροπή επανειλημμένα και για τον ρόλο των ε, κυβερνήσεων και των δράσεων, αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουμε αρκετέ υπηρεσίε ε, και οργανισμού. Έχουμε το παρατηρητήριο για την εξάρτηση και τα ναρκωτικά. Έχουμε την υπηρεσία Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που κάνει έρευνα και εξετάζει σε σχέση με τις πολιτικές που ακολουθούνται, τι γίνεται με τα κράτη-μέλη και σε σχέση με συνδυασμό, σε επαφές με εξωτερικούς οργανισμούς. Έχουμε λειτουργικές οργανώσεις, κάναμε λόγο για κάποιες από αυτές ε, σήμερα το πρωί για το Infrontex, ο κ. Ποσουτήρ που έχει την έκθεση για αυτή την υπηρεσία. Έχουμε και την αξιολόγηση σχετικά, έχουμε την Ευρωπόλ, Europol που εμπλέκεται περισσότερο και σε σχέση και με την καταπολέμηση τρομοκρατίας, ναρκωτικών, οργανωμένου εγκλήματος και διμερώς μπορούν να θεσπίζουν συμφωνίες, λειτουργικές συμφωνίες με τρίτες χώρες και οργανισμούς. Υπάρχει μια απόφαση του 2009 του Συμβουλίου ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εμπλέκεται στην αξιολόγηση αυτών των δράσεων. Έχουμε τη Eurojust επίσης για την συνεργασία στα δικαστικά θέματα όσον αφορά τις δικαστικές αρχές είναι το θέμα της ε, ε, δίωξης ε, περισσότερο. Έχουμε το θέμα της ΣΥΠΟΛ όσον αφορά την συνεργασία αστυνομικών αρχών, διασυνοριακά, επιμόρφωση, κατάρτιση. Θα έχουμε σύντομα και την υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο, για την πρακτική εφαρμογή των αρχών για το άσυλο μεταξύ κρατών μελών και συνεργασία με τις τρίτες χώρες, σε συνεργασία μέσα στα πλαίσια των υφιστάμενων συμφωνιών. Είναι κάτι για το οποίο ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο και είναι πλάκη στις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και έχουμε τώρα και την διοικητική συνιστόσα, το διοικητικό, τον οργανισμό για τα διάφορα προγράμματα IT. Ο κύριος Κουέλιο είναι υπεύθυνο το Schengen Information System, το VIS, η Eurodac και θα έχουμε και αντίστοιχη έκθεση σχετικά. Και όπως προαναφέρθηκε έχουμε και το φορέα για το συντονισμό, το όργανο, το όργανο για τις συντονιστικές δράσεις. Έχουμε και την COSI, την μόνιμη επιτροπή για την εσωτερική ασφάλεια που στοχεύει και αυτό θα το δούμε και σίγουρα για την ενίσχυση συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ Europol, Frontex, Eurojust, CPOL και το κέντρο αντιμετώπισης ε, αναγκών όλα αυτά είναι διάφορες ε, δραστηριότητες ε, και διάφοροι τρόποι με τους οποίους ε, καταβάλουν προσπάθειες αυτές οι οργανώσεις με διαφορετικές δομές. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου σίγουρα είναι διαφορετικός για κάθε μια, σε σχέση με κάθε μια από αυτές τις οργανώσεις και οργανισμούς. Έχουμε λοιπόν τα θέματα τα οποία βλέπουμε μέσα στην ομάδα μας για όλα αυτά τα σύναφη θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει δεσμευτική γνωμοδότηση από πλευράς μας για τον διορισμό ε, διευθυντών και για τους διορισμούς όσον αφορά τα συμβούλια, εκτελεστικά ή διαχειριστικά ή διοικητικά συμβούλια, διασυνδέσεις που έχει το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή μας με διάφορους από αυτούς τους φορείς, πώς διοργανώνουμε τη σχέση μας με αυτές τις επιτροπές και τα όργανα, πώς θα είμαστε σε θέση να αξιολογούμε το έργο αυτών των επιτροπών. Και όπως προηγούμενα αναφέρθηκε, αυτό είναι κάτι στο οποίο αναφερόταν και η πρόταση ψηφίσματος ε, του προηγούμενου Νοεμβρίου του Κοινοβουλίου και για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης όπου μεταξύ άλλων ζητήσαμε να υπάρξει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τα τέλη του 2010 δεν είμαι σίγουρη αν θα επιτευχθεί αυτό για ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για τη συνεργασία Europol, Eurojust να ευθυγραμμίζονται δηλαδή οι δράσεις με το Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο ζητήσαμε αναθεωρημένη εντολή για την, τον Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που θα αντιμετωπίζει και τη συνεργασία δικαστικών και αστυνομικών αρχών σε ποινικά και δικαστικά θέματα ζητήσαμε μια πρόταση ως όσον αφορά την εμπλοκή του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων στην αξιολόγηση όλων αυτών των δράσεων για την ασφάλεια και την δικαιοσύνη και τον χώρο δικαιοσύνης, ασφάλειας ε, ε, και ελευθερίας και ζητήσαμε να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες για αυτές τις υπηρεσίες και οργανισμούς ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την αξιολόγησή μας πράγμα που προβλέπεται από το ρόλο μας και να δούμε σε τακτά διαστήματα να βλέπουμε την αξιολόγηση όσον αφορά τα πολιετή προγράμματα αυτών των οργανισμών και υπηρεσιών. Ήδη έχουμε υποβάλει λοιπόν τέτοιες σχετικές προτάσεις εμείς. Ο στόχος αυτής της συζήτησης και της εγγραφής αυτού του θέματος στην ημερήσια διάταξη δεν είναι η αναζήτηση τόσο πολύ συγκεκριμένων εξειδικευμένων προτάσεων, αλλά να μπορέσουμε να δούμε πιο εξειδικευμένα και σε μελλοντικές συζητήσεις που θα έχουμε οποιασδήποτε προτάσεις που θα υποβληθούν ώστε αυτά τα θέματα να εντάσσονται καλύτερα μέσα στο πλαίσιο εργασιών και αρμοδιοτήτων της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ενώ προσβλέπουμε στη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων είναι υπηρεσίες ευρωπαϊκές αυτές και οργανισμοί ευρωπαϊκοί. Τίθεται λοιπόν το θέμα εδώ κατά πόσο και με ποιο τρόπο θα πρέπει να εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα πρέπει να διασφαλίζεται η ευρωπής εξευρωπαϊσμός, ο εξευρωπαϊσμός του έργου τους μέσα στο πλαίσιο των συνθήκων. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το ευρύτερο σκηνικό και για τα διάφορα σημεία τα οποία θα αναφύονται θα εξετάζονται μέσα από το θεσμικό όργανό μας είτε μέσω της γραμματείας είτε μέσω των πολιτικών εκπροσώπων να μπορεί να είναι και θέματα όπου κάποιοι θα θέλουν στις σημερινές και μελλοντικές συζητήσεις να λαμβάνονται κάποια πράγματα υπόψη για αυτούς τους οργανισμούς. Πρόεδρο σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν τώρα θα προσκαλέσω τον κύριο Κούκοβε, τον πρόεδρο της Κόζη, να μας προσφωνήσει, να λάβει τον λόγο. Και μετά θα ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τοποθέτησή της και θα ζητήσω ο κύριος Γιακολίνο να αναλάβει την Προεδρία για κάποια λίγα λεπτά. Κύριε Κούκοβε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μια σύντομη παρέμβαση για τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών που συμμετέχουν στην κόζη. Αναφέρομαι στην Europol, την Eurojust, την Σεπόλ και το Frontex. Στις 25 Φεβρουαρίου του 2010 το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η κόζη μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του αυτούς τους οργανισμούς και άλλους και ορίζεται με την απόφαση της 25ης Φεβρουαρίου του 2010 ότι το ΚΟΖΙ θα συντονίζει όλους αυτούς τους οργανισμούς. Συναντήθηκε, η πρώτη συνάντηση έγινε το Μάρτιο, έγιναν και άλλες δύο συνεδριάσεις υπό Ισπανική Προεδρία και καλέσαμε τις, τους τέσσερις οργανισμούς ως παρατηρητές και συμμετείχαν όλο ένα και πιο δυναμικά στις συζητήσεις ε, και στις εργασίες της ΚΟΖΗ. Ισότιμα δηλαδή με τις άλλες αντιπροσωπείες. Κατά τις τρεις συνεδριάσεις ε, της ΚΟΖΗ το θέμα της ε, συνεργασίας μεταξύ οργανισμών ετέθη στην ημερήσια διάταξη και αυτό ενισχύει το επιχείρημα για το ενδιαφέρον δηλαδή που αυτοί οι οργανισμοί έχουν για το κόσμο. Τον Απρίλιο του 2010 οι οργανισμοί παρουσίασαν ένα έγγραφο αρκετά ογκώδες στο οποίο αναφέρουν τα σημεία σύγκλησης μεταξύ τους και τα σημεία εξέτασης ε, διμερών ή πολυμερών θεμάτων. Υπάρχουν λοιπόν αρμοδιότητες που πολλές φορές επικαλύπτονται και στο έγγραφο αυτό υπάρχουν προτάσεις ούτως ώστε να διευκρινίσουμε τα πράγματα, να περιχαρακωθούν καλύτερα οι αρμοδιότητες του κάθε οργανισμού και το συζητήσαμε στις 25 Ιουνίου, στην τελευταία συνεδρίαση λοιπόν της ΚΟΖΗ. Και η Βελγική Προεδρία πρότεινε οι διευθυντές των οργανισμών να συναντιόνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει στο δεύτερο εξάμεινο του 2010 και θα την οργανώσει ένας από τους οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα η Europol. Και αυτή η συνεδρίαση των τεσσάρων διευθυντών θα γίνει και παρουσία της Προεδρίας Κόζη. Στόχος αυτών των συνεδριάσεων είναι να εγγυθούμε στην ε, κόζη τις πραγματικές εργασίες σύγκλησης των τεσσάρων οργανισμών. Ζήτησε επίσης η Βελγική Προεδρία στους οργανισμούς και βάσει των προτάσεων δηλαδή που διατύπωσαν τον Απρίλιο, να ορίσουν ένα πρόγραμμα εργασίας δηλαδή μια χρονολογική μη, απαρίθμηση των δράσεων των οργανισμών για να υλοποιήσουν τις προτάσεις που υπέβαλαν στην κόζη και η κόζη θα παρακολουθήσει από κοντά την υλοποίηση αυτών των εργασιών. Έχουμε τέσσερις συνεδριάσεις της κόζη κατά τη Βελγική Προεδρία, μία το μήνα, από το Σεπτέμβριο και μετά δηλαδή. το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών θα το έχουμε συστηματικά στις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεών μας. Και θα έχουμε και συναντήσεις στο δεύτερο εξάμεινο ε, στη συνάντηση των διευθυντών που θα γίνει από, ε, οργανωμένη από την Ευρωπόλ. Για να μπορέσουμε να έχουμε και συνεργασία μεταξύ των οργανισμών αλλά και μία συνοχή στις ε, δράσεις αυτών των οργανισμών. Είναι επίσης σαφές ότι η ΚΟΖΗ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της δεν θα διστάσει να απευθυνθεί σε αυτούς τους οργανισμούς κάθε φορά που συνεδριάζουν διότι χρειαζόμαστε τη συνεισφορά τους ούτως ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε μια στρατηγική εσωτερική ευρωπαϊκής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για ε, στενότατους συνεργάτες για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλμέιδα από την Κομισιόν. Καλημέρα σε όλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι είναι σημαντικό τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο όσον αφορά την αξιολόγηση της Europol και Eurostat με βάση τις ε, συνθήκες της Λισαβόνας θα μπορέσουν να εφαρμοστούν το άμεσο μέλλον και ήδη έχουμε ξεκινήσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αλλαγή του καταστατικού των δύο οργανισμών. Θα υπάρξει και συνάντηση αύριο του Διευθυντή μας για την ε, προετοιμασία της Europol προκειμένου να περάσει στην νομοθετική αλλαγή σύντομα. Όσον αφορά το σχέδιο δράσης, το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης ε, προβλέπει έγκριση το 2011 με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αξιολόγηση για τη Eurojust, ενώ για την Europol η ανακοίνωση αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους. Όσον αφορά τη Eurojust, το 2012 με 2013 θα καταλήξουμε κάπου γιατί πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με πολλούς εταίρους και θα πρέπει να καλύπτει θέματα όπως για παράδειγμα τις ε, ερευνητικές αρμοδιότητες ε, της Eurojust και το πώς αυτές θα εφαρμοστούν χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θέματα που μας ενδιαφέρουν είναι η σύγκριση αρμοδιότητας καθώ καθώς ε, και η αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των ομάδων της Eurojust. Τώρα, όσον αφορά τη Europol, θα υπάρξει μια ανακοίνωση για την δημοκρατική νομιμοποίηση φέτος και θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία λοιπόν για τη Europol που ελπίζουμε ότι θα καταλήξει σε έναν κανονισμό εντός του 2013. Σας υπενθυμίζω ότι το υπάρχον ε, νομικό πλαίσιο ξεκίνησε να ισχύει φέτος ε, τον Ιανουάριο. Για τον κύριο Κούκελμπεργκ να πω ότι επικροτούμε τις παρουσιάσεις των οργανισμών και της ΚΟΖΗ. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία με την Europol και την Eurojust και επίσης, όπως ε, προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης, θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε έναν τρόπο ανταλλαγής ε, πληροφοριών με την Europol και την Eurojust εντός του 2011 ή 2012. Ευχαριστώ. Έξι άτομα έχουν ζητήσει το λόγο, κυρία Ρομέρο Λόπες καταρχάς. Gracias. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε του ΚΟΖΙ για τις ε, πληροφορίες ε, που μας δώσατε. η Europol ε, και η Eurojust μπορούμε να υποθέσουμε ότι βρίσκονται τώρα σε μια νέα φάση και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να τις βοηθήσει να είναι αποτελεσματικότερες από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Θέλω λοιπόν εγώ να ρωτήσω όσον αφορά στη στρατηγική της ευρωπαϊκής ασφάλειας αν σοβαρά ε, σκεφτήκατε ποτέ σε ποιο βαθμό μπορούμε να συντονίσουμε τις υπηρεσίες πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε πολύ καλά τις δυσκολίες ε, συντονισμού αυτών των οργανισμών που διαχειρίζονται όλη την απαραίτητη πληροφορία για την καταπολέμηση του εγκλήματος και πιο συγκεκριμένα του οργανωμένου εγκλήματος Λοιπόν, ξέρουμε τα προβλήματα συντονισμού της πληροφόρησης, οπότε θέλουμε να ρωτήσουμε αν στα πλαίσια της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, να σας ρωτήσουμε κατά πόσο αυτή η ε, αυτό το τοπικό όραμα ε, θα μπορέσει να επιτευχθεί, το οποίο είναι πάρα πολύ απαραίτητο ε, θα μπορέσουμε λοιπόν εμείς ε, να προχωρήσουμε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτόν τον συντονισμό. Εμείς ε, θέτουμε, αποφασίζουμε μηχανισμούς για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, για τις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και δεν μπορούμε να συντονίσουμε τις υπηρεσίες πληροφόρησης. Προτείνω να ακούμε τις ερωτήσεις ανατρίσα και μετά να ζητάμε από τους ε, ομιλητές μας να απαντήσουν αν χρειάζεται. Ελπίζω και πάλι να έχετε αυτοπιθαρχία. Κύριε Κάνερ. Το Κοινοβούλιο για ένα χρόνο ακριβώς εξακολουθεί να βλέπει ως μυστήριο τους οργανισμούς. Όχι τόσο το τι κάνουν, αλλά για ποιον λόγο δημιουργούμε αυτούς τους οργανισμούς, ποιοι είναι οι γενικοί στόχοι τους. Μήπως μπορεί να το διευκρινίσει κάποιος αυτό. Γιατί δημιουργούνται συνεχώς νέοι οργανισμοί, ποιοι είναι η προστιθέμενη αξία τους. Επίσης, αναφέρθηκε το θέμα της ε, διαφάνειας. Εμείς στο Κοινοβούλιο πάντα ζητάμε περισσότερη διαφάνεια και περισσότερες δυνατότητες ελέγχου εκ της πλευράς μας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια είναι οι περιορισμοί στη διαφάνεια και στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και για τα εθνικά κοινοβούλια. Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες από αυτού. Ευχαριστώ ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας για τις παρουσιάσεις. Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Οι οργανισμοί είναι σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας και αυτό θα έπρεπε να φαίνεται περισσότερο στις εργασίες της ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που διαθέτει το Κοινοβούλιο για τους οργανισμούς ε, της αρμοδιότητες μας τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία δεν ήταν ιδιαίτερα καλό στα τελευταία χρόνια. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε πραγματικό νόημα το κοινοβουλευτικό μας έλεγχο. Διαφορετικά δεν κάνουμε κάτι. Και διαφορετικά τις αναλαμβάνουν άλλοι αυτούς τους οργανισμούς. Τώρα έχουμε και τον Κόζη που συμπεριλαμβάνει κάτω από την αιγίδα του όλους τους οργανισμούς και κάπου το κοινοβούλιο παραμερίζεται κάτι λυπηρό γιατί το καθήκον μας απέναντι στους πολίτες είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει καλή επίβλεψη όλων των οργανισμών. Πώς θα το επιτύχουμε αυτό θα έπρεπε τακτικώς να έχουμε σχετικά σημεία στη μερίσια διάταξη ώστε να εξασκούμε το δικαίωμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν 7 οργανισμοί που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας θα έπρεπε να τους συμπεριλαμβάνουμε στην ημερήσια διάταξη τακτικά και επίσης κάθε χρόνο να συζητάμε το πρόγραμμα εργασιών τους για το επόμενο έτος. Κάτι που δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και είναι σημαντική παράληψη. Πρέπει να ζητάμε από τους οργανισμούς να έρχονται εκ των προτέρων να μας παρουσιάζουν το σχέδιο δράσης τους για το επόμενο έτος. Αν όχι για άλλο λόγο, τουλάχιστον γιατί είμαστε και η δημοσιονομική αρχή και σε εμά θα έρθουν για να ζητήσουν κονδύλια για τον προϋπολογισμό τους. Άρα λοιπόν Αντί να συζητάμε για νούμερα κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, θα συζητάμε επί του ουσίας, δηλαδή επί των συγκεκριμένων σχεδίων που κρύβονται πίσω από αυτά τα νούμερα. Και θεωρώ ότι αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κάνει η Επιτροπή μας η ίδια, τα αναφέρω όμως για να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι και οι ομιλητές μας. Περνάω τώρα σε κάποιες παρατηρήσεις επί των ομιλιών. Καταρχάς όσον αφορά τον συντονισμό των δεδομένων, κύριε Αλμέιντα, είπατε ότι είναι πρόθεση της Επιτροπής να περάσει σε καλύτερο συντονισμό των οργανισμών κατά την επεξεργασία των δεδομένων. Στην ε, ενδιάμεση αναθεώρηση του Frontex δεν δόθηκε η δυνατότητα για κάποιο λόγο στο Frontex να επεξεργάζεται δεδομένα. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή να μας πει γιατί επέλεξε αυτή την δυνατότητα εφόσον η επεξεργασία δεδομένων θα είναι κάτι που θα απαιτηθεί σε κάθε περίπτωση, έστω και μόνο σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς. Επίσης, αρκετές αναφορές έγιναν σε αυτό το ογκώδες έγγραφο που παρουσίασαν οι οργανισμοί στην Κώση για την ε, καλύτερη συνεργασία τους. Όμως, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουμε εμεί αντίγραφο αυτό του ογκώδους εγγράφου και άρα δεν γνωρίζω πώς θα μπορέσουμε να εξασκήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας έλεγχο αν δεν έχουμε δει σημαντικά έγγραφα που πρόκειται να συζητηθούν στην Κόζη και αλλού. Παρακαλώ λοιπόν την Κόζη και ενδεχομένως την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής μας αυτό το έγγραφο. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος εργοστήσεων και πριν ζητήσω από τους κύριους Κούκομπερκ και Αλμέιντα να απαντήσουν, θα ήθελα να σας ρωτήσω Κύριε Μπουσουτήλ, έχετε συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να θέσουμε το θέμα στην ατζέντα μας, γιατί πάντα μιλάμε για μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά πώς θα το κάνουμε. Θα μπαίνει στους συντονιστές. Ναι, ιδανικά θα μπαίνει στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών προκειμένου αυτοί να καταλήξουν σε ένα συστηματικό σχέδιο για το πόσο ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των οργανισμών θα μπορούσε να ενσωματωθεί στις εργασίες της Επιτροπής μας με τακτικό τρόπο και όχι τυχαία όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να φροντίσουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Ποιος θα μιλήσει πρώτα, ο κύριος Αλμέιντα, παρακαλώ πολύ σύντομα επί των θεμάτων όπου αισθάνομαι ότι μπορώ να απαντήσω. Κάλεο, οι περισσότεροι οργανισμοί που γνωρίζω έχουν πολύ σαφείς λόγους ύπαρξης. Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνει η Europol, η Eurojust κτλ. Η Europol συλλέγει πληροφορίες για ποινικά θέματα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σεπολ καταρτίζει τους υπαλλήλους, η Frontex υπεραμείνεται των συνόρων μας από την παράνομη μετανάστευση. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν σαφείς στόχοι και σκοποί για όλους τους οργανισμούς και δεν καταλαβαίνω ακριβώς το ερώτημά σας. Όσον αφορά τη διαφάνεια, για τον οργανισμό που γνωρίζω καλύτερα, την Europol, το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή έχει πλήρη έλεγχο της, του προϋπολογισμού και έχει κάθε δικαίωμα να ζητά από την Europol να έρχεται και να εξηγεί τι κάνει. Και περνάω τώρα στο επόμενο σημείο που έθεσε ο κύριος Μπουσουτήλ που νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον μιλώντας για την δημοκρατική νομιμοποίηση της Europol. Θα ήθελα να πω το εξής. Το κοινοβούλιο και οι οργανισμοί είναι αυτοί που πρέπει να δημιουργήσουν συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφοράς που θα εφαρμόζονται κάθε φορά. Έχουμε επιτύχει πολλά όποτε έχουμε συγκεκριμένες, συγκεκριμένα ήθη που ακολουθούνται από το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια όσον αφορά τον έλεγχο αυτών των οργανισμών. Τέλος, στο ερώτημα του κυρίου Μπουσουτήλ να απαντήσω ότι ναι, είναι απόφαση της κυρίας Μάλστρομ αυτή τη στιγμή να μην δοθεί δικαίωμα στο Frontex επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τις παρεμβάσεις στα σύνορα. Αντιθέτως, η Europol έχει το δικαίωμα συλλογής προσωπικών δεδομένων για ποινικά θέματα που συμπεριλαμβάνουν και τα εγκλήματα στα εξωτερικά σύνορα. Και όντως στα πλαίσια του συντονισμού των οργανισμών θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε σε έναν τρόπο συντονισμού και κατανομής μεταξύ των τριών οργανισμών. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ κύριος Κουκουμπέρ. Θα απαντήσω φυσικά μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων μου ως πρόεδρος του ΚΟΖΗ. Ε, σας ε, ανέφερα τη σημασία που προσδίδει η ΚΟΖΗ στην ε, συνεκτικότητα και στις εργασίες των οργανισμών και αυτό δηλαδή για να απαντήσω στην κυρία Ρομέρο Λόπες για την ανταλλαγή πληροφόρησης. Το έγγραφο, το κοινό έγγραφο των τεσσάρων οργανισμών όπου αναφέρεται δηλαδή η δυνατότητα σύγκλησης και διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφόρησης που θα τη των πληροφοριών που ε, διαχειρίζονται αυτές οι τέσσερις υπηρεσίες. Αυτό το οποίο εσείς αναφέρατε όμως είναι ευρύτερο διότι προβλέπετε ένα χανές ε, ε, θέμα που έχει να κάνει γενικότερα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, με τις αστυνομίες κλπ. Μα δεν είναι το κόζι αρμόδιο για να συντονίσει, ένα, ε, για να δημιουργήσει έναν οργανισμό, να τον συντονίσει ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Εμείς αντιμετωπίσαμε το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και εσείς εδώ στο Βέλγιο. Δηλαδή πώς να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους οι διάφορες αστυνομίες και δημιουργήσαμε μια υπηρεσία που θα την ονόμαζα ως σταυροδρόμι της πληροφόρησης, είναι το ΣΕΑΝΤΕ, έτσι το ονομάζουμε εδώ στο Βέλγιο, που είναι ο Οργανισμός Συντονισμού και Ανάλυσης της Απειλής. Έχουμε δηλαδή την αστυνομία, τη δίκηση και τους εκπροσώπους ε, και τις υπηρεσίες των μυστικών ε, ε, υπηρεσιών. και μαζεύουν και αναλύουν όλες τις πληροφορίες που έχουν για τις απειλές που θα μπορούσαν να, να ενσκύψουν στο Βέλγιο και στους πολίτες του. Τώρα δεν είναι στο επιχειρησιακό σχέδιο ε, της Κόζη να κάνει τέτοια δουλειά. Δεν, είναι στο, δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητές μας. Τώρα για τον συντονισμό των διαφόρων οργανισμών και το τι θα κάνουμε ε, κατά τη Βελγική Προεδρία. Στη συνεδρίαση της ΚΟΖΗ της 25ης Ιουνίου 2010 είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω ε, στην αντιπροσωπεία της Κόζη, το πώς το βλέπει η Βελγική Προεδρία το μέλλον. Προτείναμε λοιπόν ένα πρόγραμμα που ξεπερνάει τα όρια της Βελγικής Προεδρίας και ε, θα κρατήσει κατά την περίοδο της Τρόικας. Δηλαδή καλύπτουμε και τους Ούγγρους για να έχουμε δηλαδή μία συνέχεια στις δράσεις μας. Εμείς ε, για την ε, Βελγική Προεδρία προβλέπουμε να έχουμε μια πολιτική συνέχεια με την πολιτική των Ισπανών, δηλαδή την πολιτική που ξεκίνησε από το Μάρτιο του 2010. Έχουμε πολλά ε, θέματα στα σκαριά και εμείς θα τα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε την συμβολή μας για μια εσωτερική πολιτική ε, στην Ευρώπη. Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα συζητήσουμε τα θέματα για τη στρατηγική εσωτερικής πολιτικής και ως βελγική η Προεδρία αλλά και οι Ούγγροι επίσης πρότειναν θέματα τα οποία μας καίνε και που θα θέλαμε να τα συζητήσουμε ε, στην Κόζη και είπαμε ότι θα πρέπει οι διάφορες Είπαμε οι διάφορες αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στην Κόζη, οι οργανισμοί, η Γενική Γραμματεία τον ε, το Σεπτέμβριο όταν θα συναντηθούμε για να αποφασίσουμε την ημερήσια διάταξη να μας προτείνουν και αυτοί θεματικές που τους απασχολούν. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να υποστηρίξουν αυτές τις θεματολογίες να δημιουργήσουν μεταξύ τους ε, ομάδες εργασίας ε, για να προετοιμάζουν την κόζη. Θα επιλέγονται λοιπόν τα θέματα και οι εθελοντές ε, θα... θα είναι αυτοί που θα προτείνουν λύσεις, συστάσεις στην κόζη. Έτσι θα προχωρήσουμε, δηλαδή μια προσέγγιση back down Αυτά δηλαδή. Και για να σας δώσω μια ιδέα τι θα κάνουμε στους επόμενους 6 μήνες θα συζητήσουμε για το σύμφωνο για τα ναρκωτικά θα συζητήσουμε τις 6 από τις 26 ε, λύσεις ε, για την προστασία των ε, συνόρων από την παράνομη μετανάστευση θα δημιουργήσουμε το European Crime Intelligence ε, Model έτσι όπως εγκρίθηκα και το 2005-2006 βάσει ενός ε, φιλόδοξου σχεδίου που ήταν το σχέδιο Harmony και το οποίο θα, θα συνεχίσουμε στην Βελγική Προεδρία και το οποίο στοχεύει να βρεθεί μία μεθοδολογία ούτως ώστε να οριστούν προτεραιότητες για εγγύησεις εσωτερικής ασφάλειας αντί δηλαδή να προχωράμε ε, εμπειρικά και μη πάντα επιστημονικά και καθαρά με διέστηση. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μία Ε, να έχουμε ένα εναρμονισμένο σχέδιο, μεθοδολογίες για την εσωτερική πολιτική, να μπορέσουμε δηλαδή να διαμορφώσουμε μία εικόνα για το τι εστί εσωτερική ασφάλεια, να έχουμε μία εικόνα για, τα πιο... Ε, για το τι θεωρεί ο κόσμος ε, το, ως επικίνδυνη εγκληματικότητα, να δούμε ποια φαινόμενα θα θεωρήσουμε προτεραιότητες. Θα υποστηρίξουμε την αξιολόγηση των σχεδίων COSPOL που αναθέσαμε στην Europol. Θα εγκρίνουμε έναν οδηγό για κοινέ ε, αστυνομικές επιχειρήσεις αντίστοιχα όπως γίνεται με την τελωνιακή συνεργασία. Θέλουμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εγκρίνουμε έναν οδηγό που να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη και η αστυνομικές ε, δράσεις, ε, θέλουμε να είναι κοινέ, δηλαδή να διέπονται από την ίδια λογική, από την ίδια κατοχή ε, πληροφοριών και από το ίδιο πνεύμα. Θα παρακολουθήσουμε επίσης όλες τις κοινέ δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι πάντοτε αστυνομικές αυτές οι δράσεις. Εμείς ως κόζοι θέλουμε να εγγραφούμε μέσα σε μια γενικότερη προβληματική της εσωτερικής ασφάλειας στην Ένωση ούτως ώστε να έχουμε μία ολοκληρωμένη και συνολική άποψη για την τρομοκρατία και αυτό αφορά και την αστυνομία και τη δικαιοσύνη και άλλες ε, υπηρεσίες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο ας πούμε οι υπηρεσίες ελέγχου στα σύνορα ή τα τελωνία. Αυτά σύντομα για ποια είναι τα θέματα για τους επόμενους έξι μήνες. Θα σας τα αναφέρουμε αναλυτικότερα ε, μετά τη συνεδρίαση της Κόζη στις 7 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχουμε ακόμη 7 ομιλητές. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι, κλείνω τον κατάλογο ομιλητών. Οπότε, παρακαλώ, επαναλαμβάνω, λίγη αυτοπιθαρχία και θα τελειώσουμε στα επόμενα 35 λεπτά. δε μέρα, Φλότρο και μετά Άλβαρο. δε μέρα πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σκέψεις και προβληματισμοί που συνήθως κάνω όπως πάντα. Το πρώτο θέμα είναι, εγώ συμμερίζομαι με τον Σάιμον Μπουσούτη την ιδέα που παρουσίασε ο ίδιος. Δεν υπάρχει πραγματικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αυτών των οργανισμών και επιπλέον θα πρέπει να καθοριστεί πώς θα γίνεται αυτός ο έλεγχος, διότι η κοινοτική μέθοδος που ακολουθούμε είναι κάτι εξευμενιστικό και ευγενικό. Λέει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος. Τώρα, σε σχέση με την κυρία Λάμπερτ, τον κύριο Κούκερμπεργκ και την συνάδελφο, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω σε σχέση με τον κύριο Κούκερμπεκ να μου πει γιατί δεν έχουμε το Situation Center μέσα στο ίδιο το κόσι. Θέλω να μου εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό. Γιατί σε μια δομή για την ασφάλεια δεν υπάρχει Situation Center. Δεύτερον, πιστεύω ότι από πλευρά Λάμπερτ επεξηγήθηκε τότε για τι υπηρεσίε ή οργανώσει που έχουν επιπτώσει για αυτή τη δική μα κοινοβουλευτική επιτροπή. Δεν είναι μόνο θέματα ασφάλεια και δικαιοσύνη, αλλά είναι επίση πολιτικέ ελευθερίε στην επιτροπή μα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε τον επόπτη των δεδομένων. Υπάρχει άμεση επίπτωση στην κοινοβουλευτική μα επιτροπή. Δεν είναι 7, αλλά 11. Έτσι, Σάιμον. Έλεγχο λοιπόν επ' αυτών. Από πλευρά Αλμέιδα αναφέρθηκε θεμητοποίηση, νομιμοποίηση δημοκρατική από πλευρά τη Ευρώπη. Λοιπόν, η ευρωπαϊκή νομιμοποίηση όσον αφορά την Ευρωπόλ, την Ευρωπόλ και την δομή του συνδέεται με την, τον συσχετισμό εμπιστοσύνη και πληροφόρηση με τον ε, επόπτη δεδομένων. Και αυτό γιατί, διότι είναι η ισορροπία μεταξύ πολιτικών ελευθεριών και ασφάλειας αυτό. Και είναι το κοινό πεδίο στο οποίο πάντα, πάντα το Ευρωκοινοβούλιο και κάνουμε λόγο για θέματα ασφάλειας και πρέπει να δούμε σε σχέση με την ε, εποπτεία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα από τα κλειδιά. Δεν λέω ότι πρέπει να είναι στην κόση ο επόπτης, αλλά πρέπει να ενημερώνεται πάντα τι κάνει η Κώση και να υπάρχει εμβρευστό να υπάρχουν επαφές σε εξέλιξη με την κόση, μεταξύ αυτού και της Κώση. Είναι κάτι το οποίο δεσμεύεται και συνδέεται με την νομιμοποίηση, όχι μόνο την νομιμοποίηση της Ευρωπόλ, αλλά την νομιμοποίηση των εργασιών της Κώση. Και σε σχέση με την Ευρωπόλ όλοι γνωρίζουν ότι η Ευρωπόλ έχει την ίδια τη δική της δομή, εσωτερική δομή για τον έλεγχο προσωπικών δεδομένων. Αλλά αυτό δεν επαρκεί δεν επαρκεί να υπάρχει μια εσωτερική τέτοια δομή. Αυτό που είναι αναγκαίο να γίνεται είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης στι δομέ ασφάλεια που άμεσα συνδέονται με την αναγκαία διαφάνεια που πρέπει να διασφαλίζεται. Και έτσι το είπα και το επαναλαμβάνω, ο επιθεωρητής, ο επόπτης να βρίσκεται στην ε, δομή αυτή και να βρίσκεται ρευστό σε διαρκή επαφή και να είναι πάντα ενημερωμένος για τις δραστηριότητες αυτές ε, από πλευρά των άλλων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε μέρα. Συμφωνούμε μαζί σας ε, ότι αυτό και επί χρόνια κιόλας τώρα είναι ένα θέμα μη ε, εντοπισμένου, ανεξακρίβωτου, υπτάμενου αντικειμένου. Ε, έχουμε εδώ τόσους ε, υπαλλήλους που εργάζονται μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο και πρέπει αυτά να αποσαφινιστούν. Η κυρία Φλότρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς τον πρόεδρο της ΚΟΖΕ αν ε, οι δραστηριότητες του ΚΟΖΗ χρησιμοποιούν τις εθνικές υπηρεσίες ε, και συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν ε, παράνομες πρακτικές στις υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών αποδείχθηκε για άλλη μια φορά και πρόσφατα όπου είδαμε ότι οι υπηρεσίες του τομέα αυτού αλλά και οι δικαστικές υπηρεσίες των κρατών μελών χρησιμοποιούν καταθέσεις που ελήφθηκαν μετά από βασανιστήρια, ειδικά υπό το πλαίσιο μάλλον της ε, νομοθεσίας για την τρομοκρατία. Όπως γνωρίζετε με τη συνθήκη της Λισαβόνας δεσμευόμαστε πλέον από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης υπάρχει και η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα αμφισβητηθεί αύριο μεθαύριο στο δικαστήριο στο Στρασβούργο. άλλα θέματα. Η φύλαξη των συνόρων είναι εθνική αρμοδιότητα. Όταν λοιπόν το Frontex λαμβάνει όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες, πώς το Frontex και οι υπόλοιποι οργανισμοί θα μπορέσει να εφαρμόσει τον απολογισμό των οργανισμών αυτών όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί αυτή τη στιγμή σε πολλές υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών δεν έχουν καταργηθεί οι παράνομες πρακτικές για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Δεν έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά αυτές τις πρακτικές. Μιλάμε για προστασία δεδομένων και μιλάμε πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους μηχανισμούς, τις κατάλληλες διαδικασίες για να ισχύσουν αυτά. Ευχαριστώ. Αλεξάνδρο Άλβαρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νομίζω θα μπορέσω να είμαι σύντομο, επειδή υποστηρίζω πραγματικά τι προτάσει του Σάιμον και προσβλέπω να ακούσω τι ιδέε που θα υπάρξουν όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ταυτόχρονα όμω θα ήθελα να τονίσω με ρεαλιστική προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε μια γενική τάση όσον αφορά οργανισμού και υπηρεσίε. Στην Επιτροπή Προπολογισμών το βλέπουμε αυτό που ουσιαστικά όταν καταρτίζουμε τον προϋπολογισμό των υπηρεσιών και για τον έλεγχο αυτών των υπηρεσιών υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος και κατά κάποιο τρόπο πρέπει να δημιουργηθεί δυνατότητα συμμετοχής. Θα μπορούσε ίσως να υπάρξει και ιδέα να είναι ένα μέλος του Κοινοβουλίου, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου αυτών των οργανισμών. Εξαρτάται όμως. Πώς βλέπω όμως να ακούσω τις ιδέες και τις απόψεις των συντονιστών. Μία σύντομη ερώτηση έχω μόνο προς, τον, προς Αλμέιντα. Διότι Άκουσα τις προτάσεις που υπευλήθησαν όσον αφορά την Europol. Τι θα γίνει τελικά. Θα υπάρξει κάποια αλλαγή του καθεστώτος των αξιωματούχων ε, της Europol όσον αφορά τις ασυλίες. Ε? Θα πρέπει αυτό και ευθύ εξ αρχή αναφέρθηκε θα υπάρχει ασυλία από πλευρά των υπαλλήλων αυτών. Αλλά μια και αλλάζουν τα πράγματα τώρα, αυτό θα αλλάξει ή θα συνεχίσει να ισχύει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Θέλετε να τοποθετηθείτε παρακαλώ. Καταρχάς μία μερική απάντηση στο άμεσο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Δίας Θεμέρα για την ε, ενδεχόμενη παρουσία του Σίτσεν ε, στο ΚΟΖΙ. Δεν προβλέπεται από την νομοθεσία, από την απόφαση δηλαδή του 2010, προκύπτει ότι κανένας οργανισμός ε, δεν είναι μέλος του ΚΟΣΥ, αλλά επιτρέπεται η πρόσκληση οργανισμών. Είχε προσκληθεί η ΣΕΠΟΛ και το κείμενο της απόφασης προβλέπει και ενδεχόμενη πρόσκληση σε άλλους οργανισμούς αν υπάρχει κάποιο σημείο της ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με αυτούς. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει αυτό και για τη Σίτσεν, βέβαια πάντα με καθεστώς παρατηρητή. Να απαντήσω στην κυρία Φλότχο. Το ερώτημα που θέσατε δεν ξέρω κατά πόσον αφορά ουσιαστικά την κόζη. Αναφέρεστε σε πρακτικές και αποστολές που βασίζονται σε συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των οργανισμών και τα κράτη-μέλη. Και εκεί προβλέπονται συγκεκριμένοι περιορισμοί και πάντα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα λοιπόν εξαρτώνται από τις νομικές πρακτικές των κρατών μελών. Και όπως είπατε, τα κράτη-μέλη δεν βρίσκονται όλα στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά το πώς συλλέγουν πληροφορίες οι αστυνομίες και οι υπηρεσίες πληροφοριών. Δεν θέλω εδώ να περάσω στον συγκριτικό δίκαιο, αλλά η εμπειρία μου ως Βέλγου είναι ότι στο Βέλγιο έχουμε μια νομοθεσία η οποία καλύπτει το πώς γίνεται η συλλογή δεδομένων από τους αστυνομικούς καθώς και πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Όμως αυτά δεν ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη και δεν μπορούμε βεβαίως να περάσουμε σε κάποιο είδους παγκοσμιοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Je peux και για να ολοκληρώσω, ίσως θα μπορούσα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το κοινό έγγραφο των τεσσάρων οργανισμών για τα σημεία σύγκλησης και τις δυνατότητες εναρμόνισης, συντονισμού και τα λοιπά στις καθημερινές δραστηριότητες. Το κείμενο είναι στα αγγλικά, αλλά νομίζω ότι απαντά στις ανησυχίες σας. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά, την ενισχυμένη συνεργασία ποινική και δικαστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα όχι απλώς προστατεύονται, αλλά και προωθούνται ενεργά. Μια κοινή προσέγγιση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων των οργανισμών στο χώρο της ΔΕΗ είναι λοιπόν μία υποχρεωτική προϋπόθεση. Μία καλή προσέγγιση θα έπρεπε να περιέχει συγκριτική παρακολούθηση και μηχανισμούς εκθέσεων και κατάρτισης. Και προστίθεται ότι οι οργανισμοί αυτοί θα μπορούσαν να έχουν στήριξη από τον οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος θα έπρεπε να παίζει σημαντικό ρόλο, όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Αυτά. Ευχαριστώ. Κύριο Αλμέιδα. Για να απαντήσω στην κυρία Φλότο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την Ευρωπόλ που γνωρίζω καλύτερα από τους οργανισμούς. Το μόνο θεμελιώδες δικαίωμα που μπορεί να παραβιαστεί σήμερα από την Ευρωπολ είναι η προστασία των δεδομένων. Τα κράτη-μέλη είναι δεσμευμένα να ενημερώνουν την Ευρωπολ για όλα τα εγκλήματα κλπ. Πρόκειται για ε, ε, πληροφορίες σχετικά με την εγκληματικότητα. Δεν είναι προσωπική πληροφορία. Η Ευρωπολ λοιπόν ε, μαζεύει ε, πληροφορίες από όλη την Ευρώπη, κάνει εγκληματολογική ανάλυση και αυτή την εγκληματολογική ανάλυση την ξαναστέλνει στις αστυνομίες των κρατών μελών. Το μόνο ενδυνάμει παραβιάσιμο δικαίωμα είναι η προστασία των δεδομένων. 70% από τις διατάξεις ε, που διέπουν την Ευρωπόλ είναι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των δεδομένων και υπόκεινται και σε έναν κοινό ελεγκτικό οργανισμό ο οποίος ελέγχει πολύ προσεκτικά αν γίνονται σεβαστά ή όχι αυτά τα δικαιώματα. Εμείς έχουμε ένα όριο για την αλλαγή των αρμοδιοτήτων της Ευρωπολ σύμφωνα με τη Λισαβόνα. Δεν μπορούμε εμείς ε, να δώσουμε ε, αρμοδιότητες αναγκασμού στην Ευρωπολ Εμείς ε, λοιπόν είμαστε κολλημένοι σε αυτήν την κατάσταση Δηλαδή η Ευρωπόλ για πολλά χρόνια δεν μπορεί παρά να είναι ένα κέντρο περισυλλογής ε, ε, και διάδοσης ε, πληροφοριών που αφορούν στην εγκληματικότητα. Και σε αυτή τη φάση δεν έχει, δεν, μπορούμε να δώσουμε εξουσίες, δεσμευτικές εξουσίες στην Ευρωπόλ αγγλικά. Όσον αφορά το ερώτημα για την ασυλία, θα το λάβουμε υπόψη μας. Είναι ένα από τα στοιχεία που θα λάβουμε υπόψη μας στα πλαίσια της νομοθετικής μεταρρύθμισης. Χαιρόμαστε που αύριο θα έρχουν αρκετά μέλη της Επιτροπής σας στις εγκαταστάσεις μας. Η κυρία Μάλστρομ έχει ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Europol, του Διευθυντή του Europol και την Επιτροπή ΛΥΜΠ ότι πρόκειται να γίνει μεταρρύθμιση της Europol που θα περιλαμβάνει και το θέμα της δημοκρατικής νομοποίησης από φέτος Ξεκινάμε λοιπόν αύριο με την συζήτηση όπου θα συμμετέχουν και μέλη της Επιτροπής σας και αναμένουμε την προσφορά σας όσον αφορά τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την αξιολόγηση της Europol εν ώψη της μελλοντικής μεταρρύθμισης. μου έχετε πει και ιδιωτικά ότι σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα της ασυλίας. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε. Προτείνω να πάρουμε σε ένα γύρο τους τελευταίους τέσσερις αγορητές και λαμβάνοντας υπόψη ότι πιέζει ο χρόνος, ζητώ να είστε το δυνατόν πιο σύντομοι. Για κολλήνω παρακαλώ. Θα είμαι πανσύντομος. Εγώ άκουσα με πολύ προσοχή τις ε, τοποθετήσεις που ήταν υπέρ ε, για την ενίσχυση, της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών. Η πραγματική απέτηση είναι η απόδοση της, ε, του κάθε οργανισμού. Συμφωνώ με τους ε, κυρίους Μπουσουτήλ και Ντεμέρα όταν ορίζουν μία αρχή ότι το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων, τα κονδύλια, τα μέσα και τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ε, πρέπει να ανακοινώνονται σε αυτή την Επιτροπή ούτω ώστε να μπορεί να ασκεί αυτή η Επιτροπή ένα πραγματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ε, μεγαλώνει το ενδιαφέρον για την διακίνηση ναρκωτικών. Πρέπει να βρούμε ε, τρόπους να σταματήσουμε ε, το πέρασμα των ναρκωτικών ε, που αυτή τη στιγμή περνάει, δηλαδή τη διαμετακόμιση των ναρκωτικών αυτή τη στιγμή διαμετακομίζεται από το Μαγκρέμπ. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε δυνατότητες κάθε φορά που γίνεται μία κάθε φορά που αυτές, ε, αυτοί οι οργανισμοί προχωρούν σε λήψεις μεγάλων αποφάσεων να μπορεί το κοινοβούλιο και αυτό να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο άρα να είναι και αυτό συμμέτοχο στην απόφαση. Θα έχουμε λοιπόν έτσι και ένα διαλεκτικό κίνητρο όπως έχουμε τώρα αλλά δεν θα έχουμε τίποτα αν παραμείνουμε χωρίς συνεργασία. Ευχαριστώ. Οι τελευταίοι τρει αγορητέ θα είναι Μέλο, Μπρόντ και Λάντφριντ. Παρακαλώ, η κυρία Λάντφριντ. Ο κύριο Μέλο, όχι. Μπρόντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μάλλον σαν να βασίζεται κανείς σε σχέση με τις, ε, την εργασία των οργανισμών για να διασφαλίσουμε την εσωτερική ασφάλεια. Πρέπει να δούμε τα αίτια όμως των απειλών. Πρώτα απ' όλα να σταματήσουμε τους ε, πολέμους ε, όσον αφορά τις μουσουλμανικές χώρες Αφγανιστάν και να αποφύγουμε νέους πολέμους όπως αυτό που σχεδιάζεται κατά του Ιράν. Διότι αυτοί οι πόλεμοι καλλιεργούν αντιδράσεις και βίες αντιδράσεις μεταξύ κάποιων μουσουλμάνων και στις χώρες μας και στο εξωτερικό εσωτερικό. Επίσης ε, δεν χρησιμοποιήθηκε ε, ο όρος ριζοσπαστικοποίηση και σε σχέση με τις πολιτικές ε, για τη Μέση Ανατολή όπου οι, λαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε τέτοιες αντιπαραθέσεις οι ευρωπαϊκές χώρες. Να σταματήσουμε ε, από αυτές τις χώρες που είναι πιθανοί τρομοκράτε ή εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα. Νομίζω αυτά τα προληπτικά μέτρα θα ήταν καλύτερο από το να να μπορέσουμε να συνηθίσουμε όλο και περισσότερο τις καταστατικές πολιτικές και πολιτικές περιστολής των ελευθεριών έναντι των υπόπτων. Τελευταίος η Βαρόνη Λάντφορντ. Παρακαλώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, θα μπορούσα να ρωτήσω αν η Κόζη θεωρεί την διαφθορά ως μια μίζωνα εσωτερική απειλή αφεαυτού ως θέμα για την Ευρώπη λόγω της διασύνδεσης με το οργανωμένο έγκλημα και στην ημερήσια διάταξή μας έχουμε παρουσίαση έκθεσης σε σχέση με τις διασυνδέσεις μεταξύ διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος. Συνιστώ να το εξετάσει η κόζη αυτό, διότι είναι πραγματικά ανησυχητικό το εύρος της διαφθοράς που συμπεριλαμβάνονται ακόμα και οι αστυνομικές δυνάμεις στην ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δίκτυα πορνεία και γίνεται λόγος επίσης και για πολιτικούς πάτρονες και κηδεμόνες όσον αφορά την διαφθορά, πράγμα το οποίο σημειώνεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και την επιβολή του νόμου και της δυνάμεις δίωξης. Είναι λοιπόν η διαφθορά μείζον θέμα για σας που θα έπρεπε να ήταν το εξετάζετε όπως πρέπει Κάνετε κάτι για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και να επιβληθεί ο νόμος. Και δεύτερον, για τις απειλές που αντιμετωπίζονται. Εγώ έθιξα στο, το θέμα στην Επίτροπο Μάμστρομ και στη Βελγική Προεδρία σε σχέση με την διασφάλιση της πτυχής ασφάλειας και των πληροφοριών όσον αφορά το Συμβούλιο για την ε, διάχυση στοιχείων για τη ριζοσπαστικοποίηση, συλλογή στοιχείων για την αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση. Εδώ κέντρα διαδηλωτών όπως κατά της παγκοσμιοποίησης. Δεν συμφωνώ με εκείνους που είναι αντίθετοι με την παγκοσμιοποίηση, όμως δεν θεωρώ ότι είναι απειλή. Τι γίνεται λοιπόν. Από πλευρά σας επικεντρώνεστε, επικεντρώνετε την προσοχή σας στις πραγματικές απειλές ε, κατά της ασφάλειας ε, προτού γίνουν πραγματικές απειλές και είναι δυνάμει απειλές. Οι εκόζοι και οι άλλοι συλλέγουν ή ενθαρρύνουν τη συλλογή πληροφοριών για τους διαφωνούντες και τους αντιπολιτευόμενους. Σας ευχαριστώ. Προτού καλέσω τώρα τους δύο μιλητές να ολοκληρώσουν με την τοποθέτησή τους. Πρέπει να σας πληροφορήσω και εξ ονόματος της Γραμματείας ότι η κανονική μας συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια στις 4 και 5 Οκτωβρίου θα αφοσιωθεί, θα αφιερωθεί μεταξύ άλλων και στην δημοκρατική λογοδοσία των ευρωπαϊκών οργανισμών και υπηρεσιών. Και θα έχουμε και ένα πάνελ για αυτά τον Οκτώβριο και πάλι. Κύριε Αλμίντα, σας καλώ να τοποθετηθείτε. Δεν έχετε πολλά να πείτε. Εξαιρετικό ο συμπέρασμα αυτό. Κύριε Κούκομπερ, έχετε τον λόγο. Ίσως ε, κάποιες απαντήσεις στους δύο τελευταίους ομιλητές. Καταρχάς όσον αφορά την προσέγγιση των φαινομένων ασφάλειας, ε, ε, ανασφάλειας με συγχωρείτε, και την αντιμετώπιση τους. Δεν μπορώ να σας πω και πολλά, αλλά στην ΚΟΖΗ και στους ε, υπεύθυνου για την αντιμετώπιση τους ε, μέχρι στιγμής ε, δίνεται προτεραιότητα στην καταστολή. Μιλάμε για την πολιτική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της ανασφάλειας, της έλλειψης ασφάλειας. Εκεί συμμετέχουν διάφορες φορείς, αλλά στο τέλος της αλυσίδας βλέπουμε τις δικαστικές αρχές, το ίδιο και στην αρχή αν θέλετε. Θέματα που έχουν να κάνουν με την συνοδεία, με την προστασία των ατόμων ε, και τα όλα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνουν μέτρα που θα προλαμβάνουν την, ε, τις ε, βίες ενέργειες. Και ως, τελευταίο, ως τελευταία λύση, τη καταστολή βεβαίως, μέτρα καταστολής. Τώρα όσον αφορά το αν μιλάμε για σημαντικές απειλές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσα εκ πρώτης όψεως να σας πω ναι. Όμως να σας πω ποιες είναι οι δικές μου πνευματικές ανησυχίες που θα οδηγήσουν την στη δημιουργία μιας μεθοδολογίας ολοκληρωμένης πολιτικής. Μιας μεθοδολογίας που θα μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τα εγκληματικά φαινόμενα που, στα οποία πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα που είναι τα πιο σημαντικά και πρέπει να προσέξουμε. Η διαφθορά θα μπορούσε να είναι μια τέτοια προτεραιότητα όπως επίσης ε, και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Στις 25 Ιουνίου στην τελευταία συνεδρίαση μιλήσαμε για τα εξή θέματα. Πρακτική συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ως προτεραιότητα αυτό όλα τα μέλη που ήταν στη συνεδρίαση της ΚΟΖΗ συμφώνησαν να δημιουργηθεί μία ομάδα που θα ασχοληθεί με το θέμα. Σίγουρα η διαφθορά θα μπει στην ε, ημερήσια διάταξη αυτής της ομάδας που ασχολείται με το οργανωμένο έγκλημα. Τώρα, όσον αφορά την, ε, τον ριζοσπαστισμό Μας ε, ρωτάτε αν θεωρείτε απαραίτητο να συλλέγονται πληροφορίες για τον οποιονδήποτε, για όσους μπαίνουν, για τους διαδηλωτές για παράδειγμα. Πρόκειται για πολύ ευαίσθητο θέμα. Πάντως αυτή τη στιγμή απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων για διαδηλωτές διαμαρτυρόμενους. Το σχέδιο που προετοιμάζουμε είναι να επιτρέπει στην αστυνομία να συλλέγει δεδομένα προκειμένου να μην καταλήγουν τα άτομα στην ριζοσπαστικοποίηση. Δεν μπορούμε να είμαστε τυφλοί σε ορισμένες αντιδράσεις, αλλά βεβαίως πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί και πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τον όρο. Πολύ σύντομα, κυρία Λάντφορντ. Αυτό που λέω είναι ότι το είναι κάποιος ριζοσπάστης από μόνο του. Δεν σημαίνει ότι απειλεί την ασφάλειά μας ή είναι ενδεχόμενος τρομοκράτης. Θέλω να φύγει αυτός ο όρος. Σας υπενθυμίζω ότι στην Ιταλία υπάρχει και κόμμα ριζοσπαστικό. Όταν κάποιος είναι ριζοσπάστης της απόψης του, δεν μπορεί αυτό να σημαίνει ότι είναι πιθανός τρομοκράτης. Πρέπει να είστε πολύ πιο προσεκτικοί στην ορολογία σας. Αυτός ο όρος ριζοσπαστικοποίηση είναι εξαιρετικά παραπλανητικός. Πρόεδρος, συμφωνώ απολύτως. Μας λέτε ότι δεν παρακολουθούνται οι διαδηλωτές. Δεν πάω κάθε μέρα στα διαδηλώσεις, άρα πάντα παρακολουθούνται. Υπάρχει κόσμος που βγάζει φωτογραφίες. Υπάρχουν βάσεις δεδομένων που συλλέγουν δεδομένα για τους Πιθανού ταραξίε. Υπάρχουν σε διάφορα κράτη-μέλη. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα μας. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και τους συναδέλφους που επέδειξαν την απαιτούμενη πειθαρχία. Θα επιστρέψουμε στις 3 και θα ακούσουμε την, τον Επίτροπο Ντεκούχτ που θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στην Άκτα. Ευχαριστώ.